Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben alle eine Tagesordnung bekommen. Σύντροφοι, έχετε λάβει όλη τη μέρη διάταξη. Θέλετε να αλλάξει τίποτα, όχι. Ωραία. Εγκρίθηκε σημείο 2 ανακοινώσει του Πρόεδρου. Τώρα ε, έχουμε αφενός ε, ε, συνάδελφο την ε, Σεσίλια Μόλνστρομ και οπωσδήποτε ε, και τη συνομιλία που θα έχει με τον πρόεδρο του ΠΟΕ για το Brexit και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά, όπως ξέρετε όλοι, το ΔΕΚ έλαβε μια σημαντική απόφαση για την Σιγκαπούρη που θα μας αποσχολήσει οπωσδήποτε αργότερα λεπτομερώς. Το 10 επίσης ε, έλαβε μια απόφαση για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών Stop TTIP ότι δηλαδή η τότε θέση της Κομισιόν να μην επιτρέψει αυτήν την πρωτοβουλία δεν ήταν σωστή και ε, άρα υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή η ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Κατόπιν αφού ετέθη ενισχύ η Συμφωνία Εμπορίου και η Επιτροπή συνεδρίασε στις 16 ε, Μαΐου και ο Σουηδός πρέσβης ο Ντάνιελ Μπλέκερτ εξέλεγε ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Στον ε, δε Καναδά, από ό,τι φαίνεται, ολοκληρώθηκε η διαδικασία κύρωσης ε, της ε, συνθήκης ΣΕΤΑ. Έλαβαν αποφάσεις και οι πολιτείες του Καναδά και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν θα επεκταθώ γιατί το βασικό σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα είναι η συζήτηση σε δομημένο διάλογο με την Επίτροπο την κυρία Σεσίλια Μάνστον για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το επόμενο έτος. Και βεβαίως εκεί πέρα υπάρχουν κάποια σημαντικά σημεία. Οπωσδήποτε θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο για μια εμπορική συνθήκη δεδομένου του Brexit και βεβαίως αναμένουμε και μια ξεκάθαρη θέση για μια δίκαιη εμπορική συνθήκη. Μετά οπωσδήποτε θα τεθεί το ζήτημα των σχέσεων με την Κίνα και του εξυγχρονισμού των μέσων προστασίας του εμπορίου και του νέου μεθόδου υπολογισμού προστασίας του εμπορίου που δεν θα αφορούν πλέον ε, δεν θα είναι πλέον αναχώρα και η απόφαση του ΔΕΚ για την Σιγκαπούρη οπωσδήποτε θα επηρεάσει τις ε, διαπραγματεύσεις μας με την ε, Σιγκαπούρη. Οπότε, μια σειρά καυτών θεμάτων θα έλεγα και χαίρομαι τώρα που είναι εδώ πέρα η κυρία Σεσίλια Μάνστρομ και θα μας παρουσιάσει σε 15-20 λεπτά τις προτεραιότητές της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, έχουμε έναν διαρθρωμένο διάλογο, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Σύμφωνα με την Διοργανική Συμφωνία θα πρέπει να έρχομαι εδώ πέρα συχνά για να σας ενημερώνω που βρισκόμαστε και πώς έχουν τα πράγματα. Αυτό λοιπόν θα το κάνω και βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα θέλετε που να άπτεται του διεθνούς εμπορίου. Αναφέρετε κάποια πράγματα τα οποία συνέβησαν από τότε που συναντηθήκαμε πριν από 18 μήνες όταν τέθηκε η στρατηγική εμπόριο για όλους προκειμένου να έχουμε μια πιο διαφανή βιώσιμη εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζεται σε αξίες. Από τότε εγκρίθηκε αυτή η πρωτοβουλία πολλά πράγματα συνέβησαν. Τον τελευταίο μήνα έχουμε καταρχάς την νέα διοίκηση, τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και θα πρέπει να δούμε πώς θα επηράσει τις εμπορικές μας σχέσεις. Έχουμε τις συνομιλίες για το TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες έχουν ανασταλεί επί του παρόντος ή έχουν παγώσει, αν προτιμάτε να το πούμε έτσι. Και θα προχωρήσουμε και σε νέε συνομιλίε στο μέλλον με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να αξιολογήσουμε περισσότερο τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Και προφανώ με την Αμερικανική πλευρά θα δούμε πώ μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικέ, αποδοτικέ, διατλαντικέ εμπορικέ σχέσει. Από τελευταία φορά που μιλήσαμε μέχρι σήμερα, Προέκυψε και η συγκεκριμένη πλέον εντολή για την αποχώρηση του Μένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να περιμένουμε μετά τι εκλογέ του Μένου Βασιλείου την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να δούμε στη συνέχεια πώ θα ελοποιηθεί η αποχώρηση του Μένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή η πρώτη αυτή φάση των συζητήσεων των διαπραγματεύσεων ολοκληρωθεί. Το Συμβούλιο τότε θα κρίνει πότε θα έρθει η κατάλληλη στιγμή προκειμένου για να συζητήσουμε τη μελλοντική σχέση που θα έχουμε με το Μένο Βασίλειο συμπεριλαμβανομένη εμπορική πτυχή. Έχουμε βέβαια και την ε, πιο πλήρη και σφαιρική εμπορική σχέση που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι προφανώ στην συμφωνία που έχουμε με τον Καναδά, την Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή τη στιγμή διεξάγεται η διαδικασία σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων και αυτή τη στιγμή γίνεται η τελευταία ανταλλαγή νομικών εγγράφων προκειμένου να τεθεί ενισχύ η συμφωνία αυτή το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για μια σύγχρονη συμφωνία η οποία μειώνει ήδη από την πρώτη μέρα κατά 90%, το 90% των δασμών και έχουμε και ένα νέο σύστημα δικαστικό, επενδυτικού δικαστηρίου, δηλαδή το οποίο θα ισχύει για τη συμφωνία αυτή. Αυτή τη στιγμή βέβαια το εγκρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ στρατηγικό εταίρο στο Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέρυσι είχαμε συνάψει μια συμφωνία με το Εκουαδόρ και με την Γκάνα, με την ακτή του Λεφαντοστού, καθώς επίσης και με άλλε επιμέρου χώρε τη Αφρική. Στόχο πάλι εδώ πέρα να προωθήσουμε τη διακυβέρνηση όσον αφορά το εμπόριο, να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το καθεστώ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σρι Λάνκα. Έχουμε εδώ πέρα το σύστημα GSP Plus και έχουμε μια συμφωνία ακόμα που θα συζητηθεί αύριο στην, η συμφωνία που θα συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα πρόοδος με τη Σιλάνκα, δεν δίνουμε λευκή επιταγή, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Στην τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το σύμφωνο βιωσιμότητας με το Μπαγκλαντές. Ξέρω ότι πολλοί, πολλά μέλη της Επιτροπής αυτής ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συμφωνία αυτή, ιδίως όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα στον τομέα της ένδυσης. Και έχουμε πει και στην πλευρά του Μπαγκλαντές ότι περιμένουμε και από αυτού πάρα πολύ σημαντική πρόοδο. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε σε κάθε περίπτωση να αποσύρουμε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων αν διαπιστωθεί ότι όντως δεν α, τηρούνται τα εργασιακά δικαιώματα και αυτό μάλιστα στα πλαίσια του προγράμματος όλα εκτό από τα όπλα. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανία, εξαιτίας της παρατεταμένης διένεξης καθώ επίσης και τη οικονομική επιβράδυσης και κρίση στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή έχει ζημιωθεί ιδιαίτερω. Προσπαθούμε λοιπόν εμεί από πολιτική πλευρά να δείξουμε αλληλεγγύη και να καταφέρουμε βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την αρχική φιλοδοξία τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι αύριο στην Ολομέλεια. Προσπαθούμε εδώ πέρα να προωθήσουμε προϊόντα όπως επεξεργασμένες ντομάτες, σιτάρι, καθώς επίσης και άλλα προϊόντα τα οποία από οικονομικής και πολιτικής πλευράς θα έχουν μεγάλη σημασία για την Ουκρανία. Από κοινού επίσης αποφασίσαμε για μια σειρά κανόνων όσον αφορά τα ορυκτά εκείνα τα οποία προέρχονται από εμπόλεμε ζώνε. Πάλι εδώ πέρα είχαμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώ επίση Έχουμε και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στα πλαίσια τη στρατηγική εκείνη για την καταπολέμηση των προϊόντων εκείνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα βασανιστήρια. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε πραγματικά ότι μπορούμε να οριοθετήσουμε και να διαμορφώσουμε βάσει συγκεκριμένων αξιών την παγκοσμιοποίηση και ότι μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε μεγαλύτερε ευκαιρίε ευημερία παντού στον κόσμο. Επίση, έχουμε εμπορικέ ε, συμφωνίε δεσμευτικέ ε, ιδιαίτερα φιλόδοξε, ε, οι οποίες εμπεριέχουν πτυχή για την βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς επίσης και πτυχέ όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Ξέρω ότι διήστανται πολλές φορές οι απόψει όσον αφορά την εφαρμογή των πτυχών αυτών, πάντω πιστεύουμε ότι θα καταφέρουν να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ορισμένοι ημών ζητήσετε να υπάρχουν πιο αυστηρά μέτρα, πολλές φορές ακόμα και κυρώσεις όταν οι πτυχές αυτές για τα, εμπορικ... για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα δεν εφαρμόζονται. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε επίσης ένα έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας απασχολήσει προς το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπόρου προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένε προτάσεις προς το τέλος του 2017. Για ένα-δύο χρόνια κάνουμε πολύ εντατικέ συζητήσει για την εμπορική πολιτική παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Δείχνει ότι πάρα πολλοί θέλουν τελικά να ενταχθούν στη συζήτηση αυτή. Προσπαθούμε και εμεί να ακούσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Έχουμε ανταποκριθεί σε αυτά. Έχουμε κάνει τι απαραίτητε προσαρμογέ. Έχουμε το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων που ουσιαστικά επιλύει πολλά από τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει με το προηγούμενο σύστημα ISDS της ε, επίλυσης δηλαδή διαφορών επενδυτή κράτους. Έχουμε μια πιο δεντρική προσέγγιση. Αυτή ακριβώς την προσέγγιση λοιπόν έχουμε στα πλαίσια του ΣΥΤΑ και αυτή θα προθίσουμε στη συμφωνία με το Βιετνάμ και συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Επίσης ε, έγινε μια σειρά διαβουλεύσεων όσον αφορά μια γενικότερη μεταρρύθμιση για το σύστημα αυτό, έχοντα ω απότερο στόχο να δημιουργήσουμε ένα πολυμερέ σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, στο οποίο θα συμμετέχουν πολλέ χώρε παγκοσμίω και απότερο στόχος είναι να έχουμε από ευρωπαϊκής πλευράς μια διαπραγματευτική εντολή μέχρι τα τέλη του έτους. Το εμπόριο πρέπει να είναι ελεύθερο, αλλά πρέπει να είναι και δίκαιο. Θα πρέπει να βασίζεται συγκεκριμένου κανόνες και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες και να περασπιζόμαστε το σύστημα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Βλέπουμε ότι αναδύονται κάποιες τάσεις, τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύναγγης Είχαμε ενδεχομένω κάποιε αντιπαραθέσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε ή με την Κίνα, η οποία δεν δραματίζει πάντα το ρόλο που πρέπει να δραματίζει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτέ τι πιθανέ εξελίξει. Προετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή για την υπουργική διάσκεψη. Ξέρω ότι ορισμένοι θα πάτε το Δεκέμβριο στον Πένο και επεξεργαζόμαστε και κάποια ζητήματα με άλλου εταίρου στη Γενέβη, προκειμένου να προετοιμαστούμε για την υπουργική αυτή διάσκεψη που θα λάβει η χώρα, όπω σα είπα, το Δεκέμβριο. Συστηματική και συνεχή ήταν η πρόοδο όσον αφορά τα μέσα εμπορική άμυνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε εμεί να είμαστε ανταγωνιστικοί αν πρέπει να αντιμετωπίζουμε διαρκώ αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, καθώ επίση και πρακτικέ περιβαλλοντικού και κοινωνικού dumping. Επομένω, πρέπει όλε αυτέ οι στρεβλώσει στην αγορά να τι αντιμετωπίσουμε ακολουθώντα του κανόνε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και χωρί να αποκλείουμε καμία απολύτω χώρα. Θα θέλω όμω και τη δική σα τη συμβολή για τα ζητήματα αυτά. Όπω γνωρίζετε επίση, έχουμε με ένα πολύ φιλόδοξο εμπορικό θεματολόγιο με διάφορου εταίρου. Έχουμε ολοκληρώσει εμπορικέ διαπραγματεύσει με το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη. Με το Βιετνάμ πιο συγκεκριμένα ολοκληρώνουμε τι νομικέ πτυχέ συμφωνία και θα περάσουμε από τα στη φάση τη μετάφραση. Όσον αφορά τη Σιγκαπούρη, επικαιροποιούμε το κεφάλαιο εκείνο που έχει να κάνει με την προστασία των επενδυτών. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι ο εντελεχή νομικό έλεγχο έχει ήδη γίνει και έχει ήδη μεταφραστεί η συμφωνία αυτή. Θα προσπαθήσουμε απλώ να σωματώσουμε και τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρόμαστε πάρα πολύ, την διευκρινίζω αυτή τη στιγμή, που έχουμε την απόφαση αυτού του δικαστηρίου που μα διαφωτίζει πολύ περισσότερο και αποσαφηνίζει πάρα πολύ την κατάσταση όσον αφορά τη συμφωνία αυτή και τι μελλοντικέ συμφωνίε που θα έχουμε. Θέλουμε βραχυπρόθεσμα να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Ο Πρωθυπουργό Άμπε και ο Πρόεδρο Τούσκα επιβεβαίωσαν την φιλοδοξία αυτή όταν συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στι Βρυξέλλες, καθώ επίση και στην σύνοδο του G7 στην Ιταλία. Κάνουμε κάθε το δυνατό προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία αυτή με την Ιαπωνία το συντομότερο δυνατό. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, κρεμούν κάποια δευτερεύουσα σημασία ζητήματα και θέλουμε το συντομότερο δυνατό να έχουμε την πλήρη αυτή συμφωνία με την Ιαπωνία προκειμένου να καταφέρουμε να καταργήσουμε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δασμούς που καταβάλουμε σε αιτήσια βάση, να καταφέρουμε να προωθήσουμε το εμπόριο, τις επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και να ενσωματώσουμε στη συμφωνία αυτή και ένα σύστημα εμπορικών δικαστηρίων, επενδυτικών δικαστηρίων, και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία αυτή, όπω σα είπα, το συντομότερο δυνατό. Περνάω τώρα στο Μεξικό. Πήγα στο Μεξικό πριν από δύο περίπου εβδομάδε. Συναντήθηκα εκεί πέρα με του αρμόδιου υπουργού, καθώ επίση και με εκπροσώπου κοινωνία των πολιτών, με εκπροσώπου επιχειρήσεων, εκπροσώπου του πανεπιστημιακού τομέα. Υπάρχει ένα μεγάλο επίπεδο συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού. Προσπαθούμε να συναντιόμαστε ή δυνατόν κάθε μήνα είτε σε επίσημες είτε σε άτυπες συνεδριάσεις ή μεταξύ των επισήμων συνεδριάσεων και αυτό θα συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την εμπορική αυτή συμφωνία. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Συμφωνήσαμε για τις παραμέτρους ανταλλαγή προσφορών και ελπίζω ότι θα έχουμε από την πλευρά του Μεξικού επίσης ανάλογη ανταπόκριση. Τώρα όσον αφορά το Mercosur. είχαμε εδώ πέρα μια μοναδική ευκαιρία. Επεξεργαζόμαστε και πάλι ε, την συμφωνία αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει, η οποία ελπίζουμε θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εδώ πέρα κάποια ευαίσθητα σημεία όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προϊόντα και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και με τον κύριο Χόγκεν, τον Επίτροπο τον Αρμόδιο για τη Γεωργία. Ξέρω πάντως ότι τόσο οι έμποροι όσο και τα εργοστάσια μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά και μπορεί να γίνει μια εξοικονόμηση 4 δισεκατομμύρων ευρώ όσον αφορά τους δασμούς που καταβάλουμε αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ο 13ος γύρος διαπραγματεύσεων στις συζητήσεις που έχουμε με την Κίνα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ανταλλαγή προσφορών του χρόνου Όλοι είμαστε υπέρ, φαντάζω, του λόγου που εκφώνησε στον Ταβόσο ο πρόεδρος της Κίνας. Εκφώνησε έναν πολύ θετικό επικοδομητικό λόγο. Θα πρέπει όμως τώρα η χώρα αυτή να περάσει από τα λόγια στις πράξεις και ελπίζω ότι θα καταφέρουν να διδραματίσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Έχουμε την Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα στα τέλη τη εβδομάδα και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε και εκεί πέρα να σημειώσουμε πρόοδο. Παράλληλα, συζητάμε με τέρου όπω η Ινδονησία, η Τινησία, οι Φιλιππίνε, το Μιανμάρα και ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε εκ νέου πάλι σε πραγματεύσεις με τη Μαλαισία. Και ολοκληρώσαμε την, το πεδίο εφαρμογή συμφωνία όσον αφορά την Χιλή. Πάλι θα ζητήσουμε εδώ πέρα μια διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι και ελπίζω ότι θα καταφέρει και το Συμβούλιο να κινηθεί πολύ γρήγορα προκειμένου να ξεκινήσουμε εμπορικέ διαπραγματεύσει ήδη από το φθινόπωρο. Και σα είχαμε ενημερώσει και για το ζήτημα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και θα σα ενημερώσουμε και στο μέλλον. Και ξέρετε ότι πέρυσι το Δεκέμβριο σα είπαμε ότι θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε την Ελληνική Ένωση με την Τουρκία και βρίσκονται την εξελίξη οι συζητήσεις για το ζήτημα αυτό. Καταβάλουμε προσπάθειες και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταβάλει πίεση, προσπάθειες και ασκεί πίεση αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθούν αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα, στα πλαίσια της στρατηγικής εμπόριο για όλους, προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε καλύτερα και να διαμορφώσουμε καλύτερα την παγκοσμιοποίηση, έχοντας συγκεκριμένα πρότυπα και συγκεκριμένες αρχές που δεν θα πρέπει να υποβαθμίζονται στα πλαίσια καμία συμφωνίας και αυτό έχει να κάνει με τα εργασιακά δικαιώματα, με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, Θέλουμε σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και οποιοδήποτε πρότυπο, οποιοδήποτε κανόνας όταν τροποποιείται ή όταν βελτιώνεται θα πρέπει αυτό να περνά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Θέλουμε να έχουμε πιο διαφανή και αποτελεσματική προστασία των επενδυτών με καλύτερη διάχυση πληροφοριών, με καλύτερη προστασία των ανταγωνισμού και με παράλληλη προστασία των δεδομένων. Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε τι εκθέσει και τι προτάσει μα όπω είχαμε αναλάβει και μια σχετική ευθύνη υποχρέωση στο παρελθόν. Είμαστε σε στενή επαφή με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Έγινε και ένα σχετικό διάστημα διάλογος ε, αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες και εγώ και πολλοί συνεργάτες μου έχω πάει σε πολλά κράτη-μέλη, σε πολλά εθνικά, σε όλα θα λέγαμε τα εθνικά κοινοβούλια και σε περιφερειακά κοινοβούλια επίση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε ότι το εμπόριο διδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την έκθεση προβληματισμού που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικέ εβδομάδε για την τυθάσευση, την χαλιναγώγηση τη παγκοσμιοποίηση και στα πλαίσια του εγγράφου αυτού πιστεύουμε ότι εθνικά κοινοβούλια και τα περιφερειακά κοινοβούλια, αλλά η κοινωνία των πολιτών μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν πάρα πολύ στην όλη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, ιδίω για αυτού που έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Για αυτού που δεν έχουν καταφέρει δηλαδή να εκμεταλλευτούν τα ωφέλη τη παγκοσμιοποίηση, που δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, τι κατάλληλε υποδομέ για να υποφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό που μα ενδιαφέρει πάλι είναι να έχουμε ένα ανοιχτό εμπόριο το οποίο επωφελεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τα 31 εκατομμύρια εκείνα τα οποία είναι άνεργοι. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάλι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου όλοι να μπορούν να επωφελούνται από τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές. Απότερη πεποίθησή μα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον αναδυόμενο προστατευτισμό με συγχωρείτε που βλέπουμε παντού παγκοσμίω. Προφανώ θα πρέπει να προστατεύσουμε του πολίτε μα, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργούμε νέα τύχη. Αντίθετα, θα πρέπει να δημιουργούμε γέφυρε, να διευκολύνουμε το εμπόριο και να στείλουμε το μήνυμα ότι το εμπόριο θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι όντως μπορεί να συμβάλλει και στην ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης και ότι μπορεί και η εμπορική πολιτική να συμβάλλει στην περάσπιση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δυόμιση χρόνια που μας απομένουν στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία και με εσά και με το υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να σας παρουσιάσω τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σεσίλια, για την πλήρη αυτή παρουσίαση που αφορά την εμπορική πολιτική. Για την επόμενη μία με δύο χρονιές, δυόμιση χρόνια, εν πάση περιπτώσει, πολλά, πολλά θέματα και πολλή δουλειά για την ε, Επιτροπή, αλλά και για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας. Την ευθύνη μας την παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Και επίσης παίρνουμε στα σοβαρά τις δυνατότητε που μας δίνεις για να συζητήσουμε μαζί. Έχουμε 17 λεπτά στη διάθεσή μας. Προτείνω το εξή. Κάποιο αστειάκι ακούστηκε. θα δώσω τρία λεφτά στον καθένα. Στον πρώτο γύρο θα μιλήσουν οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων και εν συνεχεία στο δεύτερο γύρο τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Κασπάρη, εξ του ΕΛΚ, έχει τρία λεφτά. Κυρία Επιτροπέ, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Τα σημαντικότερα τα έχουμε διατυπώσει βεβαίως στο εγγραφό της Επιτροπής μας, οπότε θα ήθελα να θέσω σε κάποια άλλη. Πρώτον, υπάρχει μια συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και διάβασα τη συνέντευξη του Κινέζου Προέδρου στο Νταβός. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάποια πράγματα για αυτά τα οποία ανέφερε. Είπε ότι αν κάποιος φοβάται συνεχώς να βγει στη θύελα αργά ή γρήγορα θα πνιγεί στον ωκεανό. Ε, αυτά λοιπόν αφορούν το θέμα του επενδυτικού κλίματος στην ε, Κίνα, το κατά πόσον εξακολουθεί να είναι το ίδιο ανοιχτή η κινέζικη οικονομία για επενδύσεις κατα να εξακολουθει να είναι η δική μας. Το δεύτερο είπε ο κ. Πρόεδρος, μίλησε για την ανάγκη να γίνει η οικονομική παγκοσμιοποίηση ε, πιο περιληπτική και πιο βιώσιμη. Και βεβαίως όταν μιλάμε για το αντι-dumping, ειδικά αν δούμε το θέμα της αηφορίας της ε, και της βιωσιμότητας των παγκοσμίων εμπορικών ροών, θα πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες που έχουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στον οποίο είναι μέλος και η Κίνα. Το τρίτο είπε επίση και ζήτησε μια ανοιχτή συνεργασία αμοιβαία αμοιβαία-εποφελή. Και εδώ πέρα θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, ταιριάζει αυτό με το ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν μπορούν να πουλήσουν τα αυτοκίνητα με τη δικιά τους μάρκα στην Κίνα γιατί αποκλείονται. Και να πω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ βεβαίως η καλή συνεργασία με την Κίνα, αλλά αυτό σημαίνει και τήρηση των κανόνων, ότι μπορούμε να βασιστούμε στα συμφωνημένα. Και δεύτερον, κάτι το οποίο είναι πολύ αγαπητό στην ομάδα μας, είναι το θέμα ενός πιθανού ελέγχου των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ως ΕΛΚ προτείναμε μια πρωτοβουλία νομοθετική. Θέμα μας ε, δεν είναι να κλείσουμε τις ευρωπαϊκές αγορές για τις επενδύσεις από το εξωτερικό. Χαιρόμαστε σχεδόν για όλες τις άμεσες ξένες επενδύσεις που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειαζόμαστε ε, για αυτό να υπάρχει αμοιβαιότητα, γιατί σε πολλά μέρη του κόσμου οι Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν μόνο μέρος ε, επιχειρήσεων και θα ήθελα να μου πείτε αν παρακολουθείτε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες, η κυρία Ροντρίγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσωπικές ερωτήσεις θέλω να κάνω. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρέμβασή σας. Στη δική μας ε, πολιτική ομάδα πιστεύουμε ότι η εμπορική πολιτική μας φέρνει αντιμέτωπους ε, με μια μεγάλη πρόσκληση την ε, παγκοσμιοποίηση, πώς θα τη διαμορφώσουμε, τόσο ώστε να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες, αντί να τη βλέπουν ως απειλή, να την θεωρούν ευκαιρία που δεν θα αποκλείει κανέναν. Με αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να λαμβάνουμε υπόψη την εμπορική πολιτική με όλα τα εργαλεία που διευκολύνουν την ένταξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, αλλά μια συντονισμένη δράση με την βιομηχανική πολιτική και τα, την πολιτική με των εργαλείων εμπορικής άμυνας γιατί τα εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι δημιουργούνται κινήματα εθνικιστικά, προτατευτικά, δημαγωγικά, λαϊκιστικά. Επομένως, το ερώτημα είναι πώς θα συντονίσουμε περισσότερο την πολιτική μας που θα λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία από κοινού με τα κράτη-μέλη. Επίσης, την τελευταία ολομέλεια Μιλήσαμε για μία έκθεση για την τελωνιακή εναρμόνιση. Η Κομισιόν πώς έλαβε υπόψη της τις συγκεκριμένες προτάσεις που κάναμε, ούτως ώστε να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Ε, πώς αντιμετωπίσουμε τα προϊόντα τα οποία δεν σέβονται τους κανόνες. Τι μηχανισμούς ελέγχου έχουμε, επιθεώρησης έχουμε, κυρώσεων έχουμε, ούτως ώστε τα προϊόντα τα οποία δεν σέβονται τις προϋποθέσεις να τα αντιμετωπίζουμε καταλήλως. Τρίτον, για την επόμενη Υπουργική Σύνοδο που αναφέρατε, ποιοι είναι οι στόχοι για την Κομισιόν. Μέχρι ποιο σημείο, κατά την άποψή τη, ε, πιστεύει ότι μπορούμε να φτάσουμε, να φτάσουμε σε μια συμφωνία δηλαδή που θα εγγυάται την ασφάλεια. Πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία που θα είναι δηλαδή η εξασφάλιση των πολυμερών σχέσεων, τη πολυμέρεια στο εμπόριο. Για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα στοιχεία, πώς το βλέπετε, η Κομισιόν γενικότερα, πώς βλέπει το μελλοντικό πλαίσιο των σχέσεων με, τους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις ενδείξεις που έχουμε, πρέπει να κινηθούμε έτσι πολύ προσεκτικά. Είναι πολύ λίγο αξιόπιστος ο συνομιλητής μας, είναι, θα έλεγα, πολύ αναξιόπιστος. Αυτές είναι οι γενικές ερωτήσεις. Μπορώ να μπω και στις ειδικές Α, στο δεύτερο γύρο. Έτσι, εντάξει. Στο δεύτερο γύρο θα περάσω σε πιο εξειδικευμένε ερωτήσει. Από το ECR, ο κ. Καμάλ. Ευχαριστώ, συγγνώμη. Εκπροσωπώ την Έμα Κλάρκιν, που είναι η συντονιστριά μας, αν δεν μπορούσε να έρθει. Την αντικαθιστώ, λοιπόν. Τόσο δυνατή είναι. Ε, θα μιλήσουμε για τη Σιγκαπούρη, το ξέρω μετά. Αλλά θα ήθελα να πούμε δύο λόγια, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες. Ε, πόσο καιρό θα περιμένουμε για την επικύρωση τη συμφωνίας με το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη. Δεν θέλω να πούμε σε λεπτομέρειε, είναι το επόμενο θέμα μα. Επίση, τι απόψεις έχετε για καλέ λύσει ε, για τα επενδυτικά θέματα. Ε, μιλήσατε με κάποιους εταίρους ε, μιλήσατε για το σύστημα των επενδυτικών δικαστηρίων κτλ. Τώρα, για κάτι διαφορετικό, για τις ε, διατλαντικέ σχέσει μίλησε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Για το ΤΙΖΑ, για την ε, συμφωνία δηλαδή για το εμπόριο στι. υπηρεσίε, θα κινηθούμε πιο γρήγορα και για το TTIP. Όταν ήμουν στη Ουάσιγκτον στι αρχέ του χρόνου, ε, δεν μίλησα με πολιτικού, αλλά με κάποιου υπαλλήλου κτλ. Ε, και αυτοί ακόμα είναι προσκολλημένοι στο ISDS. Ε, εμείς και ενοχλούνται από το γεγονός ότι εμεί περάσαμε στην, ε, στο σύστημα ε, των επενδυτικών δικαστηρίων. Ε, εσύ έχετε και εσείς αυτέ τι ενδείξεις ότι είναι κολλημένοι οι Αμερικάνοι εκεί στο ISDS, το Μηχανισμό επίλυση δηλαδή Διαφορών ε, Επενδυτών κράτου για το Μερκοσούρ και την πρόσβαση για τα γεωργικά προϊόντα και τα πρότυπα για τα τρόφιμα. Ε, τα σκάνδαλα για το, για το κρέας ε, δημιούργησε αβεβαιότητα στη διαπραγμάτευση ε, και για το SPS οι άλλοι, οι εταίροι μας ας πούμε τι λένε. Καθυστερούνται οι διαπραγματεύσεις εξαιτία αυτού. Ελπίζω να, συμπεριφερθούμε, να συμπεριφερθούμε ως ενήλικες και να κινηθούμε. Επίσης για τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωση με την Τουρκία. Πώς θα προχωρήσουμε δεδομένων το, του πολιτικού πλαισίου. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτή η εναρμόνιση δεδομένη πολιτικής κατάστασης. Υπάρχουν κάποιοι από εμά που θέλουμε πολλές πολιτικές, ε, εμπορικές συγγνώμη, συμφωνίες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και τα πολιτικά δεδομένα. Η άποψή σας ποια είναι. Ευχαριστώ από την ε, Άλντε, του τους Σα Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, που χαρτιγραφήσατε τόσα πολλά θέματα, επί των οποίων θα εγγύψει η Κομισιόν και όλοι μα. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά και οι γεωγραφικές περιοχές που καλύπτατε, καθώς και τα οριζόντια θέματα. Ε, Παραδείγματο χάρη δυτή χρήση, ε, καταπολέμηση των εργαλείων που χρησιμοποιείται για βασανιστήρια, ε, μεταλλεύματα από εμπόλεμες περιοχές. Ε, όλα αυτά δείχνουν πώς ε, οι εμπορικοί κανόνες μπορούν να μας βοηθήσουν και σε αυτά τα θέματα. Επίσης, για τους κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο είπατε ότι η προστασία των δεδομένων και ο προστατευτισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό εδώ στην Ευρώπη εμείς να δείξουμε πώς αυτοί οι κανόνες μπορούν να διαμορφωθούν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες, καθώς οι Αμερικάνοι μάλιστα είτε ψάχνονται ακόμα είτε χαλαρώνουν τις προσπάθειές τους και μια και υπάρχουν πολλές αλλαγές, θα ήθελα να μου πείτε τι εμπειρίες αποκομίσατε από τη Ουάσιγκτον και αν μπορείτε να μας μιλήσετε λιγάκι για το αν το Συμβούλιο, από ό,τι ξέρετε, θεωρεί, από ό,τι ακούω εγώ στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον, ότι υπάρχει μια έτσι, νέα ορμή ε, για την Ευρώπη. Ή έχει αλλάξει τίποτα. Η Ιαπωνία, το Μεξικό και άλλες χώρες αλλάζουν τη στάση τους, γιατί επηρεάζονται από τη στάση των Αμερικανών. Πώς πιστεύουν ότι μπορούν να διαμορφωθούν οι συγκεκριμένες πολιτικές με καλύτερη εντολή κτλ. Γιατί πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όσο μας επιτρέπει ο πιο δημοσκρίκος μας πέρα από την, πολιτική κατάσταση στο Συμβούλιο, μα μας πείτε λιγάκι περισσότερα πράγματα για την απόφαση για τη Σιγκαπούρη και τα επόμενα βήματα, καθώς και τα μέσα υπεράσπισης του εμπορίου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό εδώ να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ελπίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορμή, τη νέα ορμή, για να παίξουμε ηγετικό ρόλο στο να έχουμε ένα εμπόριο με κανόνες και διμερός και πολυμερός. Και αυτό πρέπει να το προτάξουμε στις επαφές μας με τις τρίτες χώρες. Ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μια που η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο να πω το εξή. Έχουμε εδώ πέρα μια μεγάλη κατσαρόλα στην οποία έχουμε πάρα πολλά συστατικά και αναγνωρίζω πράγματι ότι υπάρχει μια μεγάλη ατζέντα που σας απασχολεί και έχει όλες τις μελλοντικές προκλήσεις. Είπατε ότι το θέμα δεν είναι μόνο το ελεύθερο εμπόριο αλλά το δίκαιο εμπόριο και συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ακριβώς η πτυχή αυτή του δίκαιου εμπορίου. Αν μιλάμε για ενίσχυση του πολυμεριούς εμπορίου, μιλάμε για διαφορετικά πράγματα και δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Και αυτό βεβαίως αφορά και την 11η Υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες για τους οποίους το Γερμανικό Υπουργείο έχει πει ότι ακόμα και το να γίνει θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και αυτό έρχομαι σε τρία-τέσσερα ερωτήματα. Το πρόγραμμα εργασία πάντα πρέπει νομίζω να έχουμε κατά νου την σχέση με τους αναπτυξιακούς ε, στόχους που αφορούν το περιβάλλον, τα κοινωνικά και την αναπτυξιακή πολιτική. Δηλαδή, οι στόχοι αυτοί του ΟΗΕ θα πρέπει να αποτελέσουν ένα μέτρο σύγκρισης για την περαιτέρω εξέλιξη της στρατηγικής αυτής. Οπότε, είπατε ότι η εντολή για πρέπει να διαπραγματευτείτε την έντολη για ένα πολυμερές εμπορικό δικαστήριο. Το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί αυτή η εντολή και αν έχουμε και εμείς την δυνατότητα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επηρεάσουμε και να επηρεάσουμε ουσιαστικά για να καταλήξουμε πραγματικά σε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη ε, διάφορες πτυχές της επενδυτικής πολιτικής μεταξύ των οποίων και τις υποχρεώσεις των επενδυτών ε, π.χ. δεδομένων, την ρύθμιση και το θέμα του ψηφιακού εμπορίου και τέλος για ένα ακόμα θέμα, είπα. Με ενδιαφέρει εδώ πέρα πώς η Κομισιόν με βάση την παλαιά εντολή της ε, TTIP θα διαπραγματευτεί τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Πώς θα έχει προσεχώς η διατλαντική εμπορική σχέση. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους, κυρία Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Μόλις βγήκα από μία συζήτηση όπου είχαμε και έναν υπάλληλό σας από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ατιμορρησία στο Μεξικό μέσω του εξυγχρονισμού της συνολικής συμφωνίας. Υπήρχαν διάφοροι ειδικοί που ενδιαφέρονταν να δω αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα που σχετίζεται με το σύστημα δικαιοσύνης, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας, τα βασανιστήρια κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο των συμφωνιών νέας γενιάς. Δεύτερη ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση του ΕΛΚ και θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρόταση αυτή για τις πηγές χρηματοδότησης που είναι παραδείγματο χάρη βρώμικο χρήμα, διαφθορά κτλ. Και το επόμενο ερώτημα αφορά την χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης όπως λέγεται. Έχω γράψει τρία σημεία εκεί πέρα. Υπάρχουν τρία σημεία που λένε πως η Κομισιόν ε, είναι έτοιμη να προτείνει κάποιες δεσμευτικές ε, περιβαλλοντικές και εργασιακές προδιαγραφές και η Κομισιόν λέει όταν όμως οι εταιρείε δεν παίρνουν στα σοβαρά τις υποχρεώσεις τους για το περιβάλλον και τα εργασιακά θα πρέπει να λογοδοτούν. Θα καταλήξει κάπου αυτή η φράση σας εδώ πέρα. Και για το EFTD η κυρία Μπέγγιαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας. Κάποιες ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, η απόφαση, η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θεωρούσε ουσιαστικά μη αποδεκτή την πρωτοβουλία των πολιτών Stop TTIP, ε, που ξέρετε ότι είχε συγκεντρώσει πάρα πολλές υπογραφές από πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος λοιπόν εμείς τώρα θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να ληφθεί βέβαια υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον. Πώς προτίθεστε εσείς να προχωρήσετε λοιπόν, πώς την πράξη θα δώσετε συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρώτον αυτό, δεύτερον. Σε σχέση με την εμπορική πολιτική και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να μας ενημερώσετε λίγο όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς και ιδίως όσον αφορά τις ε, εισαγωγές ε, κρέατος, όπως ακριβώς προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Τρίτον, επιστρέφουμε εμείς, ορισμένα μέλη της Επιτροπής δηλαδή, το Φινικέλιο. Επιστρέφουμε από μία αποστολή στην Ινδονησία. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει κάποιες ε, διαπραγματεύσεις και θα θέλαμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τι προβλέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το φινικέλαιο. Και τελευταία τώρα ερώτηση όσον αφορά την αναθεώρηση της Γεωργικής Συμφωνίας με το Μαρόκο. Χθε εγκρίθηκε η διαπραγματευτική εντολή. Εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα κάποιο αντίγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίσουμε και εμείς πότε θα μπορούσαμε να έχουμε διαθέσιμο αυτό, το, αυτή την εντολή διαπραγματευτική. Ο κύριος Φερόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ σήμερα σε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση. Εσείς είστε ο υπέρμαχος ή υπέρμαχος μάλλον των ελεύθερων συναλλαγών στις Βρυξέλλες. Μια ερώτηση λοιπόν θα ήθελα να σας κάνω ιδιαίτερα ειλικρινή σε σχέση με τις συζητήσεις αυτές. Θέλετε να δώσετε νέα όθηση, είπατε νέα πνοή στις εμπορικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε απογοητευτεί όμως λίγο με την νέα Αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλτ Τραμπ που προωθεί περισσότερο τον προστατευτισμό, τους δασμούς και το ερώτημά μου είναι λίγο διαφορετικό βέβαια. Εσείς λέτε ότι θέλετε να αναζαγωνίσετε την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με ποιον ακριβώς θα το κάνετε αυτό. Να σας δώσω εγώ κάποιες ιδέες. Προτείνατε διεύρυνση δεσμολογική με την Τουρκία. Είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό να το συζητήσουμε εδώ πέρα, προκειμένου να συμπεριλάβουμε και τα γεωργικά προϊόντα και τι υπηρεσίε. Ενδεχομένω να μην γνωρίζετε όμω ότι δεν έχουμε καλά καλάβγια από το ρωσικό εμπάρκο και είχαμε πριν από δύο μέρες την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στις Βερσαλίες στη Γαλλία και το ζήτημα αυτό δεν ετέθη. Επομένως, ποια θα είναι η δική σας η προσέγγιση όσον αφορά κατά αναλογία την Τουρκία, η οποία μπορεί και αυτή να απειλήσει με τη σειρά της στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αυτή η δασμολογική συμφωνία λοιπόν με την Τουρκία, την οποία προτείνετε εσεί, έχει μια έντονη πολιτική πτυχή που δημιουργεί προβλήματα και επίσης ε, δημιουργεί και ορισμένου φόβους και αμφιβολίε σε ορισμένε πολιτικές ομάδες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη ερώτηση προς την Επίτροπο λοιπόν, η ε, δασμολογική αυτή ε, ένωση με την Τουρκία θεωρήθηκε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως ένα προήμιο, αν θέλετε, μια εισαγωγή στην ε, διεύρυνση προς τη χώρα αυτή. Ξεκίνησε το 2005 αυτή η διαδικασία, αυτή τη στιγμή έχει παγώσει από ό,τι καταλαβαίνω, που βρισκόμαστε λοιπόν με τη δασμολογική αυτή ένωση και όσον αφορά την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε συμπερίληψη των δύο αυτών πτυχών στις γεωργικές συμφωνίες, γιατί ε, οι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλουν να γνωρίζουν τελικά τι θα προκύψει από τη συμφωνία αυτή. Γιατί η δεσμολογική αυτή ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας θα απειλήσει χρηματοοικονομικά τους ε, Ευρωπαίους γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε τρόπον την αν τους καθησυχάσουμε. Σας ευχαριστώ. Δέκα λεφτά τώρα έχεις εσύ, Σεσίλια, να απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Κάποιες από τις ερωτήσεις σας ήταν κοινέ ε, για τις πολιτείες, Φερρυπίν. Κύριε Κασπάρη, χάζει για την Κίνα. Ο πρόεδρος της Κίνας δεν θα προσκληθεί στη Σύνοδο αλλά ο Πρωθυπουργό θα έρθει. Παρ' όλα αυτά θα θέσω αυτά τα θέματα, γιατί ε, και εμάς μας άρεσε η ομιλία εντυπωσιαστήκαμε από την ομιλία του, αλλά όχι από την πραγματικότητα της Κινίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πραγματικότητα και είναι δύσκολο να επενδύσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι ε, στην Κίνα. Ε, υπάρχουν πολλές διακρίσεις, δεν υπάρχει διαφάνεια, ε, ε, κρατικές ενισχύσεις, ε, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, μακρός, μακρύς ο κατάλογος και πρέπει να τα δούμε. Το εμπόριο με την Κίνα θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Είναι πολύ εύκολο να κάνουν εμπόριο οι Κινέζοι εδώ και γενικά είναι καλό πράγμα αυτό, παρότι υπάρχουν ε, επιφυλάξει, θα πρέπει και εμείς να μπορούμε να κάνουμε εμπόριο εκεί. Και ο σκοπός μια τέτοια επενδυτική ε, συμφωνία είναι να υπάρξει ισότητα. Ελπίζω να συμφωνήσουμε με τους ε, Κίνου, Κινέζους για την ανταλλαγή των προσφορών, ώστε να προχωρήσουμε και σε αυτό το θέμα. Για την ε, εξέταση των ξένων γράφων θα το συζητήσουμε στην Κομισιόν είναι δύσκολο το θέμα, γιατί έχει νομικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσει και θα πρέπει να το δούμε σωστά και προσεκτικά. Ε, θα γίνει σύντομα μία ε, σύνοδος με τους επιτρόπους για να το συζητήσουμε και εκεί θα εντάξω και το δικό σας έγγραφο. Για την παγκοσμιοποίηση. Πολλά από τα θέματα στο έγγραφο ήταν μια απόπειρα για να δημιουργηθεί μια στρατηγική για την παγκοσμιοποίηση. Ήταν ένα έγγραφο εργασία. Δεν έκανε συγκεκριμένε προτάσει ε, και δόθηκε στα κράτη-μέλη στη γενική συζήτηση που θα κάνουμε για την. Θα το δώσουμε μάλλον, θα κάνουμε για την Ευρώπη. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση τη εμπορική πολιτική, που είναι ένα τμήμα τη παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει η διαφθορτική, περιφερειακή, κοινωνική πολιτική, πώ θα χρησιμοποιήσουμε τα κοινά μα κονδύλια με πιο έξυπνο τρόπο, πιο γρήγορο τρόπο, πώ μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει και ένα δίκτυο προστασία για τα άτομα τα οποία είναι ξεχασμένοι ε, τη παγκοσμιοποίηση, που ε, υφίστανται τι ε, αρνητικέ συνέπειε. Τώρα που βγαίνουμε από την οικονομική κρίση, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε να κάνουμε κάτι και για αυτού. Συμφωνώ ε, ότι η φόρο διαφυγή είναι τεράστιο θέμα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, το κάναμε και στο πλαίσιο του G20. Ναι, αυτό το έγγραφο θα οδηγήσει σε μια πιο συνεκτική στρατηγική, ελπίζω όχι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τι μπορούν να κάνουν πολύ πιο συγκεκριμένα τα κρατημέλια αλλά και με καλύτερη, καλύτερο συντονισμό. Buenos Aires. Ο στόχο είναι να ενισχύσουμε το σύστημα του ΠΟΕ. Φυσικά, πολλέ χώρε, παρότι δεν συμφωνούμε μαζί του για τα πάντα, συμφωνούμε παρόλα αυτά ότι ο ΠΟΕ έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και θα τον ενισχύσουμε. Συνεργαζόμαστε με πολλέ χώρε, στην Γενέβη, με του πρέσβει του, ε, προτάσεις παραδείγματος χάρη για τις ε, αλληλευτικές επιδοτήσεις, ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαφάνεια για τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χώρια στήριξη, θα συζητηθεί και αυτό. Θα γίνει μια υπουργική την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι, στο πλαίσιο του ΟΣΑ, όπου πολλοί υπουργοί θα συζητήσουν ένα απόγευμα τις τα προπαρασκευαστικά του Μπένος Άιρες Και ελπίζω να προχωρήσουμε λιγάκι. Βεβαίω μπορώ να επανέλθω και να σας ε, εξηγήσω. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές ερωτήσεις από πολλούς από εσά. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο νομίζω. Το TTIP αναφέρθηκε αλλά δεν συζητήθηκε λεπτομερώς. Ο υπουργό Εμπορίου ε, των ΗΠΑ χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να το δει. Εάν ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, Πώ θα προχωρήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, τότε δεν χρειαζόμαστε εντολή. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό ή πιο περιορισμένο, ίσω χρειαζόμαστε μια φρέσκη εντολή. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τι προποθέσει. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, επιβάλλουν πολλά προστατευτικά μέτρα, α πούμε, στην αγορά κρατικών προμηθειών, στι ε, ναυτιλιακέ υπηρεσίε, ε, που αλλάζει λιγάκι τι συνθήκε. Θα πρέπει να ξέρουμε. Αν λοιπόν ξαναρχίσουμε τι διαπραγματεύσει, από πού θα τι πιάσουμε, υπό ποιε συνθήκε. Ε, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε. Και βεβαίω χρειαζόμαστε κάποιο θεματολόγιο για τις διατλαντικές μας επαφές. Ε, υπάρχει και το θέμα του ΤΙΖΑ. Ε, προς το παρόν δεν μας έχουν απαντήσει οι Αμερικανοί. Ε, η κυρία Ρέντινγκ ε, το παρακολουθεί. Ε, Πολλέ χώρε μα λένε τι να κάνουμε, προσπαθήσουμε να ξαναρχίσουμε τι ε, διαπραγματεύσει, γιατί είχαν προχωρήσει πάρα πολύ. Και το ίδιο συμβαίνει και για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Ε, αλλά ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν επιθυμεί πλέον πολυμερεί ε, εμπορικέ συμφωνίε. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Δεν συζήτησα μέχρι στιγμής με τους πολιτικούς ε, το ISDS ή το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις από τους Αμερικανούς, αλλά οι επικρίσεις για το παλιό σύστημα ε, τις ασκούσαν και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο, το παλιό σύστημα για δηλαδή το ISDS. Επομένω υπάρχει άνοιγμα για τη Σιγκαπούρη. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση, θα γίνει μια τεχνική συνεδρίαση για να σα ενημερώσω. Ε, το καλό είναι όμω ότι δίνει μια σαφήνεια. Λέει ότι είναι ε, για την προστασία των επενδυτών λοιπά έχουμε επιμερισμένη ε, ευθύνη. Ε, είναι σαφήνει αυτό. τώρα πώς θα επηρεαστούν οι μελλοντικέ συμφωνίε με τη Σιγκαπούρη και οι υπόλοιπε μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε θα δούμε. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Δεν σημαίνει... Τι σημαίνει αυτό, τι διαιρούμε, τι εμπορικέ συμφωνίε στο μέλλον. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Να προχωρήσουμε με, το, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια διαδικασία επικύρωση. Θα πρέπει να βγάλουμε έξω τι επενδύσει θα πρέπει να το δούμε αναπερίπτωση. Υπάρχουν πολλές επιλογές για να προχωρήσουμε. Ελπίζω να βρούμε μία λύση, ούτω ώστε να κάνουμε εμπορικέ συμφωνίες και επενδυτικές συμφωνίες και να μπορούμε με κάποιο έτσι, λογικό τρόπο να τις επικυρώνουμε. Ούτω ώστε να μην παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και περιμένουν και οι εταίροι μας ε, αιώνια, αλλά να υπάρχει και το δημοκρατικό στοιχείο εντός τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε τα κρατημέλη αυτό το θέμα. Και μαζί σας εννοείται. Για το Μερκοσούρ ο κ. Ανδριου ε, την επόμενη εβδομάδα με το σκάνδαλο για το κρέας πήγε εκεί, στη Βραζιλία. Ε, και είπε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει η Βραζιλία. Είναι παράλυση τη αυτή με το Μερκοσούρ. Το κεφάλαιο του SPS είναι ένα από τα κεφάλαια που θα πρέπει να το δούμε έντονα στις διαπραγματεύσεις του Μερκοσούρ, των φυτογενομικών δηλαδή θεμάτων. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Πρέπει να το δούμε και ανεξάρτητα από το σκάνδαλο του κρέατος. Τουρκία. Είναι μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπάρξει ανανέωση αυτή τη παλιά ε, τελωνιακή συμφωνία που περιορίζεται μόνο στα βιομηχανικά προϊόντα. Η νέα συμφωνία λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβει όχι μόνο τη γεωργία αλλά και τις ε, κρατικές προμήθειες, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Το Συμβούλιο το ζήτησε τρεις φορές στα συμπεράσματά του, μετά από την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, να υπάρξει αυτή η ανανέωση της συμφωνίας, διότι συνειδητοποιούμε τις συζητήσεις που κάνουμε με την Τουρκία, που είναι δύσκολες συζητήσεις, ούτως ή άλλως είναι δύσκολος εταίρος και η πολιτική της Τουρκίας μας απασχολεί υπό πολλές έννοιες. Είναι όμως μια ευκαιρία να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε κάτι που πιστεύουμε και η ΜΕΝ και η ΔΕ ότι είναι υποφελέ. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή υπάρξει εντολή και ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, ω συνήθω θα είμαστε πάρα πολύ απέναντι στο, ανοιχτοί απέναντι στο Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να εξηγήσουμε πώ λειτουργεί το πράγμα. Και κύριε Φεγό, ναι, είμαι υπέρμαχο των ε, ελεύθερων συναλλαγών στην Ένωση. Είναι τμήμα του, της δουλειά μου. Φυσικά είμαι απογοητευμένη από πολλά προστατευτικά μέτρα που έχει λάβει η Αμερικανική κυβέρνηση. Κύριε Σάρκ. Ρωτήσατε κάποια πράγματα, νομίζω απάντησα, αλλά νομίζω ότι κάποια από τα γεγονότα στην Ουάσιγκτον, δηλαδή η απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να φύγει από την TPP όπως υποσχέθηκε, αυτό σημαίνει ότι οι άλλες 11 χώρες απογοητεύτηκαν πολύ και όλες ήρθαν σε επαφή μαζί μας και μας είπαν να επιταχύνουμε τις υφιστάμενες διαπραγματεύσεις ή να κάνουμε το επόμενο βήμα κτλ. Παστράφηκαν στην Ευρώπη και μας ζήτησαν επίσης να υπερασπιστούμε το πολυμερές ε, σύστημα και νομίζω ότι έτσι άλλαξε κάπως η διάθεση στο Συμβούλιο, ότι τώρα δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ένας νέος τρόπος εμπορικών συμφωνιών που θα είναι δίκαιες, αμοιβαία υποφελής, να κερδίζουν και οι δύο πλευρές και είμαστε σε επαφή με ε, πολλές χώρες. Οπότε υπάρχει φιλοδοξία όσον αφορά το εμπόριο και κάποια περισσότερη αισιοδοξία σε σχέση με πριν από έξι μήνες. Δίκαιο εμπόριο, συμφωνώ κύριε Σόλτς σε πολλές ε, χώρες, ε, π.χ. στη Λατινική Αμερική, προσπαθούμε να τους εκπαιδεύσουμε σε διάφορα θέματα δίκαιου εμπορίου. Θα γίνει μια ανακαίνιση φέτος και για το βραβείο αυτό, ε, δίκαιου εμπορίου. Για το πολυμερές δικαστήριο βεβαίως γράφουμε μια αξιολόγηση αντικτή που είμαστε σε επαφή με άλλες χώρες, γιατί δεν είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, είναι μια διεθνής πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε εμείς τους όρους, αλλά βεβαίως μπορούμε να ζητήσουμε μια ευρωπαϊκή εντολή για το ποια είναι τα σημαντικά σημεία. Και νομίζω ότι θα το αποφασίσει αυτό η Κομισιόν αυτό το τέλος του έτους και θα ζητήσει από το Συμβούλιο κάτι και βεβαίως μπορούμε να το συζητήσουμε το φθινόπωρο όταν θα ξέρουμε περισσότερα ε, ακριβώς για να ενταχθεί στην διαδικασία. Η κυρία Χάουτα, αλλά το θέμα της ατιμορρησίας στο Μεξικό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολλά προβλήματα σχετίζονται με αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί όμως να λυθεί με μια εμπορική συμφωνία, αλλά βεβαίως η διαπραγματεύσει με το Μεξικό είναι στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης και τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα, να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί για το φινικέλαιο. Κύριε Πικέ, υπάρχει ένας φάκελος ο οποίος ετοιμάζεται και οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχουν βεβαίως αναλάβει τον ε, βασικό ρόλο ε, και εμείς συνεισφέρουμε αλλά ίσως μπορείτε να ρωτήσετε αυτούς για περισσότερες λεπτομέρειες. Για τις διαπραγματευτικές οδηγίες για το Μαρόκο, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και Τελωνιακής Ένωσης επίσης είναι αρμόδια. Όχι εμείς, αλλά οπωσδήποτε θα σας ενημερώσουμε. Και θα σεβαστούμε οπωσδήποτε το... την απόφαση του δικαστηρίου, όπως πάντα. Με, κοιτάτε, ναι, κύριε Πρόεδρε, ε, είχα πολλές ερωτήσεις όμως. Τέλος. Κύριε Μπεγκίν, ε, το γνωρίζουμε το ζήτημα το οποίο θέσατε. Και ο κύριος Χόγκαν είναι ήδη σε επαφή με τους ε, συναδέλφους ε, του κλάδου της Γεωργίας στη ΣΥΠΑ. Ελπίζουμε να βρούμε μία λύση, αλλά δεν έχουμε ακόμα καταλήξει. Αυτά νομίζω. Σας ευχαριστούμε. Τώρα έχουμε 14 άτομα που έχουν ζητήσει τον λόγο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μισή λεπτό ο καθένας. Λοιπόν, 1,5 λεπτό. Ωραία, ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που συμμετέχετε σε αυτόν τον διάλογο. Φυσικά θα έχετε πολλή δουλειά. Μία ερώτηση για το χρονισμό στην πολιτική που είναι σημαντικός. Καταρχάς για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ. Είμαι και ο εισηγητής. Αλλά ισχύει και για την Συμφωνία με το Μεξικό και τη Χιλή. Μας είπατε ότι θέλετε να τελειώσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2017. Σας ρωτάω εάν έχετε συνέστηση του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο καθυστερεί τουλάχιστον ένα χρόνο για να χτενίσει τα κείμενα, για να, να κάνει την αναθεώρηση από τους νομομαθείς, ε, γλωσσομαθείς μάλλον κτλ. Ε, μην ξεχνάτε ότι η συμφωνία με το Μερκοσούρ έχει ευαίσθητα σημεία και για τους δύο πλευρές. Επίσης, ε, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο, ε, εμπόριο αξίας ενός δισεκατομμυρίου με την ε, Ιαπωνία. Επίσης, μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας εμείς για να μπορέσουμε να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες και αν θα προλάβουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία και κάτι άλλο. Ε, μπορείτε να κάνετε εσείς κάτι, να κινητοποιήσετε όλους τους ανθρώπινους πόρους σας, ώστε να τα καταφέρουμε να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες στη δική μας κοινοβουλευτική θητεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επανέλθω στην απόφαση του δικαστηρίου για την Σιγκαπούρη. Εγώ πριν από δύο χρόνια έλεγα ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τι δύο συμφωνίε την επενδυτική από τα αγαθά και υπηρεσίε. Δεδομένη απόφαση και του ότι απορρίφθηκε το κομμάτι περί αγαθών και υπηρεσιών, μήπω θα πρέπει να έρθει το κομμάτι αυτό στο Κοινοβούλιο και να κυρωθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό και στο μέλλον, νομίζω για να απαντήσω στην ερώτησή σα θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστέ συμφωνίε επενδύσεων και ελευθέρου εμπορίου και τον... Ε, πώς λέγονται? συμφωνίε σύνδεσης, σε μπάση περιπτώσει. Νομίζω πρέπει να έρθουν χωριστά οι συμφωνίες της Σιγκαπούρης. Δεύτερον, Το δικαστήριο τώρα είπε ξεκάθαρα ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, άρα πρέπει να έχει και αποκλειστική αρμοδιότητα για την έγκριση το Κοινοβούλιο και όχι άλλα κοινοβούλια. Θα αντισταθείτε στις προσπάθειες του Συμβουλίου να εισαχθούν νέοι τομείς ε, στις εντολές μελλοντικών ε, συμφωνιών ε, ελευθέρου εμπορίου για να το εμποδίσει αυτό. Μας έχει δώσει μια ευκαιρία το δικαστήριο και πρέπει να τα αρπάξουμε από τα μαλλιά. Σας ευχαριστώ. Αν Μαρή Μινέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και κυρία Μανωστρών που ήρθατε να μιλήσετε για την εμπορική πολιτική από τις 16 Μαΐου γνωρίζουμε την απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αρμοδιότητα των κρατών μελών και είναι κρίμα ε, το ότι ε, κάθε φορά το δικαστήριο λέει ότι οποιαδήποτε επιδιαιτησία θα πρέπει να πηγαίνει στα κράτη-μέλη από τις 10 ε, Μαΐου και το είπε η κυρία Τετσιάνα Μαΐ, το είπε η κυρία ε, γνωρίζουμε ότι κακώς απέρριψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρωτοβουλία πολιτών για το Stop Σέτα και τη με 3,5 εκατομμύρια υπογραφές. Δεν έπρεπε να την έχει παραμερίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην δημοκρατική συζήτηση. Θέλω λοιπόν να μάθω τι θα κάνετε με αυτές τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Λέτε ότι δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων και θα πρέπει να έρχεται εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει χαμηλότερη συμμετοχή και λιγότερες αρμοδιότητες. Θα μπορούσατε όμως από την άλλη να λάβετε υπόψη τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες των πολιτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεστε στις δικές τους ανησυχίες. Βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος να ε, υπάρχουν τελείως διαφορετικές συμφωνίες από αυτές τις οποίες θα θέλετε, αλλά ως δημοκράτης δεν νομίζω να έχετε καμία αντίρρηση. Σας ευχαριστώ. Έρχομαι κατευθείαν από την ομάδα παρακολούθησης της Δυτικής Σαχάρας και πρέπει να σας πω ότι ε, συγκλονίστηκα για το ότι χτες ε, δόθηκε η εντολή για νέες διαπραγματεύσεις και σήμερα έχουμε την ομάδα παρακολούθησης. Δεν είναι ε, διαφάνεια αυτή, η διαφάνεια για την οποία μας μιλάτε συνεχώς, ούτε ο απαιτούμενος σεβασμός της Κομισιόν απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, στα συγκεκριμένα θέματα. Άκουσα ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον όγκο του εμπορίου της Δυτικής Σαχάρας. Ε, πώς μπορείτε τότε να διαπραγματεύεστε. Φαντάζεστε να είχατε διαπραγματευτεί την ΣΕΤΑ γιατί ε, χωρίς να γνωρίζετε τι ακριβώς διαπραγματεύεστε. Το δεύτερο. Με ποιον θα διαπραγματευτείτε. Άκουσα, ε, δεν υπόθηκε ρητός, ότι πιθανώς ε, θα μιλήσετε με, τις, με τους ντόπιου εκπροσώπους των κατοίκων. Δεν είπε το δικαστήριο. Το δικαστήριο απέτησε να μιλήσετε με τον πληθυσμό, τους κατοίκους της Σαχάρας. Πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να διαπραγματευτείτε με τις δυνάμεις κατοχής για το τι ε, θα κάνει ο κατεχόμενος πληθυσμός. Ευχαριστώ. Κύριος Βίζας. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Σε σχέση με τη ΣΕΤΑ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακχόν, ζήτησε να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για να μετρήσει και να αξιολογήσει την ε, συνθήκη ΣΕΤΑ. Εσείς τι άποψη έχετε. Μπορεί αυτό να καθυστερήσει την έγκριση της ε, ΣΕΤΑ. Και επίσης ε, ο David Μάρτσας έκανε μία ερώτηση για τις μεικτές συνθήκες. Τελικά τα κράτη-μέλη μπορεί να έχουν τον τελευταίο λόγο για πολλά θέματα. Ε, και μπορεί να καθυστερήσουν ή να παρεμποδίσουν την ε, υπογραφή μιας συμφωνίας. Ε, είναι πολύ λογικό αυτό που υπόθηκε. Να, να περιοριστούμε δηλαδή στα θέματα τα οποία είναι αποκλειστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εμπορικά θέματα δηλαδή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ε, θα αναφερόταν όλο και περισσότερο στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών στη βιώσιμη ανάπτυξη στα κοινωνικά εργασιακά πρότυπα. Έχετε αρχίσει να επεξεργάζεστε την αρχική αυτή ιδέα και είχαμε πει ότι ενδεχομένω να πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση βάσει κυρώσεων στην Ευρώπη και υπάρχει πλειοψηφία υπέρ αυτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι περισσότεροι εμπορικοί μα εταίροι φαίνεται ότι έχουν ήδη εγκρίνει μια τέτοια προσέγγιση. Δείτε λίγο τι διατάξει ε, για το TPP, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση πραγματικά να ανασχηματίσει εντελώ την προσέγγιση τη όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντο και να προβλέπει πραγματικά κυρώσει για παραβίαση αυτών των προτύπων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπαν ο κύριο Φίσα και ο David Μάρτιν όσον αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Και όπω είπαν και οι συνάδελφοι από την ΓΚΟΕ, θεωρώ ότι πραγματικά εδώ πέρα εκπροσωπούμε, εκπροσωπούμε του πολίτε εδώ πέρα. Και εντάξει, αν κάποιο θεωρεί ότι δεν εκπροσωπεί του πολίτε, μάλλον θα πρέπει να αποχωρήσει και από το Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε σε έναν διεξοδικό κατάλογο με πάρα πολλού εμπορικού εταίρου. Ενδεχομένω να έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερε εμπορικέ διαπραγματεύσει από ό,τι είχαμε ποτέ στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα όμω που τίθεται είναι το ακόλουθο. Όλο και περισσότερο προκύπτει το εξή ζήτημα. Πετυχαίνουμε πραγματικά αυτό το οποίο θέλουμε μέσω των συμφώνιων αυτών. Το θέμα των δασμών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μείωση λοιπόν των δασμών, η κατάργηση των δασμών το εμπόριο στη συνέχεια, αλλά βλέπουμε στη συνέχεια ότι υπάρχουν διατάξεις που δεν χρησιμοποιούνται τελικά από τους εταίρους. Νότιος Κορέας, για παράδειγμα, 65% μόνο, στο 1078% στο Μεξικό μόνο 52%. Μόνο ένα 52% των επιχειρήσεων, των παραγόντων χρησιμοποιούν τελικά τις ευνοϊκές διατάξεις που εμείς συμπεριλαμβάνουμε στις συμφωνίες αυτές, ενώ οι περισσότεροι επικεντρώνονται τελικά στους κανόνες καταγωγής των προϊόντων. Ειλικρινά λοιπόν δεν βλέπω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο για το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένες εμπορικές αυτές συμφωνίες στο μέλλον. Κάποιες συμφωνίες πρόσφατες όπως αυτή του Βιετνάμ έχουν κάνει τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων λιγότερο ευέλικτους σε σχέση με τους κανόνες που είχαμε στο παρελθόν. Πώς ακριβώς λοιπόν θα μεταρρυθμίσουμε τους κανόνες προέλευσης των προϊόντων γιατί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν διευκολύνουμε καθόλου τελικά το εμπόριο στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Κυρία Μάλμστρομ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ερώτηση έχω. Τώρα με την απόφαση του ΔΕΚ είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες για τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά δεν είναι σαφές το εάν είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο το νέο αυτό σύστημα εμπορικών δικαστηρίων. και βέβαια αυτό ανεξαρτήτως με το τι θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Μετά για το Brexit ενεργοποιήθηκε το άρθρο 50, έχουμε συμφωνίες που ισχύουν και περιλαμβάνουν και τη Μεγάλη Βρετανία. Τι σημαίνει αυτό, πώς το βλέπετε και κάτι άλλο για την Τουρκία. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα γίνει με τον εξυγχρονισμό της ε, Τελωνιακής Ένωσης και πότε θα εγκριθεί μια εντολή. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντινγκ. Μία ε, πρόταση για την ορολογία. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για ελεύθερο εμπόριο, αλλά θα πρέπει να μιλάμε πια για δίκαιο εμπόριο. Αυτό θα ήταν και μια απάντηση σε πολλούς από τους πολίτες που θέτουν ε, ερωτήματα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο προστατευτισμός όλο και αυξάνεται σε πολλές χώρες εταίρους και θα στην κατάλληλη στιγμή να κάνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή επίθεση για να απαντήσουμε σε αυτές τις τάσεις. Το τι Φερρυπίν. Τα περισσότερα μέλη τα οποία διαπραγματεύονται την ΤΙΖΑ είναι συμβαλόμενα μέρη του TTIP. Και σχεδόν με όλα αυτά τα μέρη έχουμε διμερεί σχέσει με όλε αυτέ τις χώρες. Επομένως θα ήταν προς το συμφέρον μας και προς το δικό τους να προχωρήσουμε. Και χρήσιμο θα ήταν να πάρουμε μια πρωτοβουλία για να κάνουμε κάτι. Πολλά δε μάλλον που οι πολυμερείς σχέσεις, η πολυμέρεια μπορεί να είναι ο προθάλαμος της, του multilateralism. επενδύσεις. Η πρόταση που παρουσίασε και μας είπε ο κύριος Κασπάρη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε ένα εργαλείο ελέγχου των ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη. Γιατί το πράγμα είναι τελείως μπερδεμένο και αντί να έχουμε μια σαφήνεια δεν έχουμε σε καμία περίπτωση. Και αντί να, και για να απαντήσουμε και στο, τις τάσεις του προστατευτισμού, γιατί να μην έχουμε και μια ευρωπαϊκή έτσι, πράξη, αυτό θα διευκρίνιζε και τη θέση μα. Μαρία Αρένα. Σα ευχαριστώ. Στον αφορά την απόφαση για τη Σιγκαπούρη, το δικαστήριο μας είπε ότι δεν αναφέρθηκε στη συμβατότητα, αλλά στη συνύπαρξη διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Μήπως και πάλι εδώ πέρα υπάρχει ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά το ζήτημα της συμβατότητας το είπε το ίδιο το δικαστήριο στα πλαίσια της γνωμοδότησής του και αυτό γύρει ένα θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι συμβαίνει με το ζήτημα της συμβατότητας. Δεύτερον, όσον αφορά τα μέσα εμπορική άμυνας, επεξεργάζεστε όπως μας είπατε διάφορα μέτρα κατά του ντάμπινγκ και διάφορα άλλα μέσα εμπορική άμυνας, θεωρώ ότι υπάρχουν εδώ πέρα δύο αρχές που ουσιαστικά υπονομεύουν την αρμοδιότητα που έχουμε για να καταπολεμούμε κατά του ντάμπινγκ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, πολλές φορές τα ίδια τα ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν μας επιτρέπουν τελικά να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα εμπορικής άμυνας. Υπάρχουν συγκεκριμένε πρακτικές dumping όταν υπάρχει συγκεκριμένη στρέβλωση τη αγορά. Πρέπει λοιπόν να δούμε εμεί τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή και ποια μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και δεύτερον, μία συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά την χαλιβουργία, τον κλάδο της χαλιβουργίας σε πάρα πολλές χώρες. Κάποιες έρευνες δείξουν ότι υφίσταται ντάμπινγκ και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα γιατί λέει ότι προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού λαού τελικά και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Αν πάρουμε όμως την περίπτωση της Ρωσίας, της Ουκρανίας όσον αφορά τη χαλιβουργία θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε τι πιστεύετε για το ζήτημα αυτό. Τέλος, όσον αφορά μια πρωτοβουλία που θα πρέπει εσείς να αναβάλλετε για την δέους επιμέλεια, ειδήσω όσον αφορά την υπόθεση και την ένδυση. Υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πραγματικά δείχνουν ότι θα πρέπει επιτέλους εσείς να λάβετε δεσμευτικά μέτρα δέους επιμέλειας όπως ακριβώς έχουμε πάρει για τα ορυκτά τα οποία προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες. Ο Πιάντρο Τασίλβα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αναφέρατε την ε, Ιαπωνία και είπατε ότι αποτελεί πρωταρχική σας προτεραιότητα όσον αφορά το εμπορικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είμαι μόνιμος συζητητής για την Ιαπωνία. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για την ανακοίνωση αυτή. Είπατε ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ ο φάκελος. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να γνωρίζω αν μπορείτε ήδη από σήμερα να μας περιγράψετε κάπως την συμφωνία όσο έχει αυτή τη στιγμή. Είναι μια προοδευτική συμφωνία τελικά. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε στα πλαίσια τη συμφωνία αυτή. Ε, μια δεσμευτική πτυχή, ένα δεσμευτικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και πώς θα αντιμετωπίσετε την αντίσταση της ιαπωνικής πλευράς όσον αφορά το σύστημα ISDS. Θα λέγατε ότι ο μηχανισμός αυτός επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους τελικά είναι καλύτερος από το να έχουμε ένα κακό σύστημα επίλυσης διαφορών. Θα έπρεπε να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής με την Ιαπωνία. Πρόεδρος, είμαι Ροντρίγκερς, Τελευταίο ομιλητή. Που θα μα εκφράσει προσωπικέ τη πια απόψει όχι τη ομάδα. Με μικρόφωνο κατά καλύτερα. καλύτερα. Δύο συγκεκριμένε ερωτήσει. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι ε, Φιλιππίνες που έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ. Ε, Μόλι ε, παρουσίασε μια έκθεση το Human Rights Watch για αυτό το θέμα. Η Κομισιόν σκέφτεται να αναδιατυπώσει το σύστημα γενικευμένα προτιμήσεων πλάς ε, απέναντι στις Φιλιππίνες και τι μέτρα μπορεί να λάβει ούτως ώστε να διορθωθεί αυτή η φρικτή κατάσταση. Δεύτερο ερώτημα. Λογικά η εμπορική πολιτική άλλαξε, βελτιώθηκε και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, συμφωνίες όμως, σε σχέση με συμφωνίες που έχουν υπογραφεί παλιά, μήπως θα μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιον ευέλικτο μηχανισμό ε, εξυγχρονισμού των παλιών συμφωνιών, ούτω ώστε να μπορέσουμε τις πιο καινοτόμε πτυχές που αφορούν ας πούμε, τη βιώσιμη ανάπτυξη να τις εντάξουμε σε αυτές τις παλιές ε, συμφωνίες και να μην ε, ξανακάνουμε όλη την περίπλοκη αυτή διαδικασία, αλλά που θα μας επιτρέπει παράλληλα να προχωρήσουμε και να εξυγχρονίσουμε και αυτές τις παλιές συμφωνίες που δεν έχουν αυτά τα στοιχεία. Και εγώ τώρα κάποια σχόλια. Το Brexit. Η Τερέζα Μέη μόλις δήλωσε είπε ότι ε, το να μην υπάρχει συμφωνία δεν είναι καλύτερο από την κακή συμφωνία. Ποια είναι η γνώμη σας. Υπάρχει προετοιμασία για το no deal, για το καμία συμφωνία. Ποια θα ήταν η καλή συμφωνία επίσης. Για να έχουμε έτσι και ένα, μια πηξίδα ένα μπούσουλα. Ετοιμάζεται επίσης μια λύση για την ε, διαδικασία επικύρωσης των, διαδικασιών, των συμφωνιών με τρίτες χώρες. Θα αντιγράφουμε, κάθε φορά θα αντιγράφουμε ας πούμε, τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με άλλες χώρες ε, απλό copy-paste δηλαδή. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλαφράνκα, το Μάιο του 2019 θα γίνουν οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εμπορικές συμφωνίες ε, είναι χρονοβόρες. Δεν προσπαθούμε να τις ε, καθυστερήσουμε. Προσπαθούμε να τις επιταχύνουμε όσο μπορούμε. Φέτος εστιάζουμε και δίνουμε όλους τους πόρους, ούτως ώστε το, η συμφωνία με την Ιαπωνία, το Μεξικό και το Μερκοσούρ ε, να ολοκληρωθούν. Η μετάφραση παίρνει χρόνο. Ε, η νομογλωσσική επεξεργασία επίσης. Θα διαπραγματευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει αυτή η κοινοβουλευτική θητεία να κάνει πολλά Δεν σα λέω να δουλεύετε μέχρι τελευταία στιγμή, α πούμε λίγο πριν τι εκλογέ, αλλά τουλάχιστον να μην σταματήσετε τον Ιανουάριο, κύριε Μάρτιν. Ε, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Θα ήταν μια επιλογή αυτή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι σήμερα, ναι, αυτή είναι η επιλογή να διαιρέσουμε τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Θα μπορούσε στο μέλλον να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Χρειάζεται όμω να το εξετάσουμε με τα κρατη Και αν αυτή είναι και η άποψη του Κοινοβουλίου, η δική σας μόνο ως ε, εισηγητή, ε, καλό θα ήταν να τη λάβουμε υπόψη μας. Το δικαστήριο. Πολύ κάνετε αυτήν την ερώτηση. Το δικαστήριο ξεκαθάρισε τα πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ε, συμφωνιών ελευθερών εμπορίου είναι αποκλειστική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Δηλαδή η επικύρωση στα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον δημοκρατικό τρόπο ε, με το θέμα. Δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε τα εθνικά κοινοβούλια. Κάνουμε πολλέ συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Ε, όλη η διαδικασία γύρω από τη ΣΕΤΑ μα έκανε να σκεφτούμε. Ε, πρέπει να εμπλέξουμε τα εθνικά κοινοβούλια. Και όχι μόνο τελευταία στιγμή και μεμονωμένα, αλλά από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πολλού τρόπου για να το κάνουμε. Μπορούμε να του πούμε σήμερα αποφασίσαμε για την εντολή για να διαπραγματευτούμε συμφωνία με την χή χώρα. Η Κομισιόν θα ξεκινήσει αύριο. Ας δημιουργήσουμε την Επιτροπή, όπου ο, Επιτροπο, ο Υπουργός σας, ας πούμε, θα σας ενημερώνει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Είναι ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων. Δεν είναι ευθύνη τη ε, Κομισιόν. Εμεί παίζουμε απλώ το ρόλο μα και θα το κάνουμε. Δεν είναι αντιδημοκρατικό το να επικυρώνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι μπορούμε να επικυρώνουμε και συμφωνίε με δημοκρατικό τρόπο, διεξοδικά, αλλά χωρί να, να, χρειάζεται χρειάζεται χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τελικά δεν έχουν κανένα νόημα αυτέ οι συμφωνίε. Το πώς θα το κάνουμε ακριβώ ε, στο μέλλον αυτό όμω, δώστε μα λίγο περισσότερο χρόνο. Θα την τεχνική συζήτηση σήμερα το απόγευμα και εγώ θα είμαι στη διάθεσή σα ε, λίγο αργότερα για την πιο πολιτική συζήτηση. Η Κομισιόν προτείνει εντολέ, κύριε Μάρτιν, αλλά δεν εγγυάται την, τελική έκβαση στο Συμβούλιο. Εμεί προσπαθούμε να παίξουμε το ρόλο μα απλώ. Κύριε Μίνα, και ζητώ συγγνώμη κύριε Μπεγκίν που δεν σα απάντησα. Έχουμε λάβει Έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για το TTIP, που δεν λέει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί. Ήταν λάθος της Κομισιόν να το καταγράψει αυτό και η Κομισιόν θα πρέπει να το διορθώσει τώρα. Ήταν μόνο το θέμα της καταχώρησης που ήταν λάθος. Δεν είπε τίποτα για το περιεχόμενο. Κύριε Μπούχνερ, για το Μαρόκο ναι, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όπως είπε και το δικαστήριο, για να ενσωματώσουμε και τους, τον λαό τη υποσαχάριας Αφρικής. Δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Η υπηρεσία εξωτερική δράση ψάχνει να βρει διάφορου τρόπου για να το κάνει. Αποφασίστηκε χθε μόλι, είναι υπό την ευθύνη τη υπηρεσία εξωτερική δράση και το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται για αυτό το θέμα. Κύριε Φίσα, διάβασα στι εφημερίδε ότι ο κύριος Μακχόν θέλει να δημιουργήσει αυτή την ομάδα εργασίας. Δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Μακχόν για αυτό το θέμα, ούτε με την κυβέρνησή του. Θέλει να δει δηλαδή τι επίπτωση θα έχει στη Γαλλία πριν το επικυρώσει το Γαλλικό Κοινοβούλιο, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Λογική πρόταση. Δεν σημαίνει ότι η προσωρινή εφαρμογή που θα ξεκινήσει σύντομα είναι να αμφιβόλο, τίθεται να Είναι μια εσωτερική γαλλική διαδικασία για να εμπλακεί το κοινοβούλιο και να, να είναι σίγουροι οι Γάλλοι ότι υπάρχει διαφάνεια, η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Αναφέρθηκα. Α, κυρία έχει φύγει. Τέλο πάντων, δεν απαντώ ερώτηση αυτή, λοιπόν. Απαντήσω, τέλο πάντων. Ανέφερε ήδη στην αρχή τη παρέμβασή μου ότι επεξεργαζόμαστε ένα έγγραφο για τη βιώσιμη ανάπτυξη η πτυχή αυτή, τα κεφάλαια τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεσμευτικά. Το ότι δεν υπάρχουν κυρώσει πολλέ φορέ δεν σημαίνει ότι τα κεφάλαια αυτά δεν είναι δεσμευτικά. Θα προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιε συναλλακτικέ, θα ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά και εναπόκειται στη συνέχεια στα κράτη-μέλη και σε εσά και στι μη κυβερνητικέ οργανώσει και στην κοινωνία των πολιτών να συμβάλλουν στην όλη συζήτηση. Κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να έχουμε και κυρώσει. Επίσης, ένα ακόμα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο ετέθη στο, στην προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου είχε να κάνει με την εφαρμογή. Πολλές φορές έχουμε σε θεωρητικό επίπεδο καταπληκτικές συμφωνίες, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν καλά στην πράξη. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε καλύτερα πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά συμφωνίες αυτές και πώς μπορούν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συχνά επιχειρήσεις εκείνες που δεν έχουν πρόσβαση στα ωφέλη των συμφωνιών εμπορικών συναλλαγών. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να βελτιώσουμε και τα συστήματα πληροφορικής όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής και σύντομα, λίγο αργότερα φέτος τουλάχιστον, θα υπάρχει και μια έκθεση όσον αφορά τη συγκεκριμένη εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών και βέβαια περιμένουμε και τις δικέ σας προτάσεις. Τώρα η επόμενη ερώτηση. Δεν ζητήσαμε από το δικαστήριο να γνωμοδοτήσει για το σύστημα των επενδυτικών δικαστηρίων. Θέλαμε να δούμε που υπάρχουν παράλληλες συντρέχουσες αρμοδιότητες. Είμαστε πεπισμένοι ότι το νέο αυτό σύστημα συνάδει και συμμορφώνεται με το νοσιακό δίκαιο. Ξέρω ότι η βελγική κυβέρνηση θα, θα θέσει στο δικαστήριο το ζήτημα αυτό. Ήδη για κάτι τέτοιο και εμείς θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις όλες διαδικασίες. Είμαστε πεπισμένοι πάντως ότι το σύστημα το οποίο προτείνουμε εμείς συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο. Τώρα, όσον αφορά το Brexit, και απαντώ εδώ πέρα και στην ερώτηση του Προέδρου. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε εμπορικέ συμφωνίε, όταν αποχωρήσει όμω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποχωρήσει και από τι ευρωπαϊκέ εμπορικέ συμφωνίε. Μπορεί στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο να συνάψει εκ νέου συμφωνίε με του εξωτερικού εταίρου Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό να απόκειται σε αυτό. Τώρα, πότε θα έχουμε την επικαιροποίηση της Ελληνική Ένωσης με την Τουρκία. Αυτό θα γίνει όταν θα έχουμε και μια διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα. Και θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια δύο χρόνια περίπου για να, διαπραγμα... για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις. Κυρία Ρέντινγκ τώρα, ναι όντως, προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε επίθεση κατά του προστατευτισμού με αυτό το πολύ φιλόδοξο θεματολόγιο, καθώς επίσης και με όλες αυτές τις διμερείς, πλειονομερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις που προωθούμε, όπως είπα πριν από λίγο υπάρχουν πάρα πολλέ χώρες που συμμετέχουν στη ΤΙΣΑ και μας ρωτάνε αν μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί μας με ή και χωρί τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και βέβαια θα είναι πολύ κρίμα να μην ευοδοθεί τελικά η συμφωνία αυτή μόνο και μόνο επειδή θα υποχωρήσουν αποχωρήσουν, με συγχωρείτε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Όσον αφορά τώρα την παρακολούθηση των επενδύσεων. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να εξετάσουμε εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Θα ξεκινήσει πάντω η συζήτηση αυτή και έχω ήδη και το έγγραφο του ΕΛΚ στα χέρια μου και θα επανέλθουμε σίγουρα στο ζήτημα αυτό όσον αφορά τη διαδικασία παρακολούθηση και επιτήρηση Απάντησα στο ζήτημα τη ε, συμβατότητα. Τώρα, Όσον αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας, νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά και σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις θελήσαμε να δούμε πώς κατά περίπτωση μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο εμπορικής άμυνας στο οποίο αναφερθήκατε. Και πάλι εδώ πέρα όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την δέους επιμέλεια και τον τομέα της ένδυσης. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο ισχύει για τα ορυκτά τα οποία προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες. Θα ήταν πολύ πολύπλοκο αυτό. Έχουμε τις κατευθύνες γραμμές του ΟΣΑ για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Δεν νομίζω όμω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να συνάδει απόλυτα με το σύστημα το οποίο έχουμε θεσπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα ορυκτά από εμπόλεμε ζώνες. Ναι. Η διαπραγματεύση στην Ιαπωνία θα είναι σαν την ΣΕΤΑ, θα έχει κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη και το σύστημα των επενδυτικών δικαστηρίων. Πράγματι δεν το έχουμε λύσει ακόμα με την Ιαπωνία. Φιλιππίνες, ναι. Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Ήμουν εκεί πριν από δύο μήνες για την διασκέψη του Αζίαν. Το έθεσα το θέμα με τους εταίρους μας ότι ανισχούμε πολύ για κάποια ζητήματα, τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, ε, τις εξοδικαστικές εκτελέσεις και κάποια άλλα θέματα και τους προειδοποίησα ότι βεβαίως ε, ε, μπορεί να υπάρξει μια αναστολή του καθιστώτος προτιμήσεων. Θα το ξαναδούμε το φθινόπωρο, αλλά η κατάσταση είναι πολύ ενισχυτική πράγματι. δεν υπάρχει τώρα τρόπος να εξυγχρονιστούν γρήγορα οι παλές ε, συμφωνίες. Χρειαζόμαστε εντολή από το Συμβούλιο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, θα είναι εξαιρετικά τυχές. Οι όροι ε, του Brexit ευτυχώς ε, είναι κάτι το οποίο αφορά τους ανωτέρους μου. Ελπίζω λοιπόν ο κύριος Μπαρνιέ και άλλοι να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν μια καλή συμφωνία. Ηνωμένο Βασίλειο είναι φίλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ελπίζω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε καλές μελλοντικέ σχέσεις. Οι εμπορικέ διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν ακόμα, είναι νωρί Νομίζω θα ήταν ατυχές ε, εάν δεν καταλήγαμε σε κάποια συμφωνία και ας μην απελπιζόμαστε ακόμα. Αυτά νομίζω. Ωραιότατα. 29 και ένα λεπτό νωρίτερα. Ωραιότατα, σας ευχαριστούμε Σεσίλια και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε διάφορα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα. Την απόφαση του Δικαστηρίου για την Συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Επιτέλους, λοιπόν, ξεκαθάρισε το θέμα των αρμοδιοτήτων το εάν είναι μια μεικτή συμφωνία ή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιο κομμάτι ανήκει πού. Κάτι το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Εμείς, ε, το Κοινοβούλιο δηλαδή πάντα, ήμασταν ε, στις ε, συζητήσεις βλεπόμενοι. Απευθύναμε και μια επιστολή στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Τώρα βεβαίως το συναρπαστικό ερώτημα είναι τι θα βγει από αυτό και τι θα κάνουμε με τις ε, συμφωνίες. Ο David Μάρτιν πρότεινε να σπάσει η συμφωνία. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα κάνουμε με την απόφαση του ΔΕΚ. Και εδώ πέρα υπάρχουν τέσσερα άτομα λοιπόν που θα κάνουν μια μικρή εισαγωγή στο θέμα Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που έχουμε εδώ τον αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, στον οποίο δίνω μέσα στον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι στις 16 Μαΐου, η 16η Μαΐου ήταν σημαντική ημέρα γιατί εξέδωσε την ε, γνωμοδότησή του το Δικαστήριο για τις Αρμοδιότητες για τη Συμφωνία Ελευθερίου με την Σιγκαπούρη. Ε, η απόφαση λήφθη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου και ξεκαθάρισε επιτέλους τα πράγματα για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες για το μέλλον των εμπορικών συμφωνιών. Και μάλιστα ε, εμείς ως Κομισιόν χαρήκαμε γιατί απάντησε ξεκάθαρα στο ερώτημα που θέσαμε το οποίο δεν αφορούσε την συμβατότητα με την δική μας συνθήκη, αλλά το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Ποιο κομμάτι δηλαδή της συμφωνίας είναι αποκλειστικά για την Ένωση και ποιο δεν είναι. Και θα ήθελα να πω ότι όταν πήγαμε στο δικαστήριο και θέσαμε το ερώτημα αυτό, χαρήκαμε που μας στήριξε το Κοινοβούλιο και Μάλιστα, σε όλες τις προτάσεις της ε, Κομισιόν μας βοήθησε το Κοινοβουλίο. 25 κράτη-μέλη επίσης παρενέβησαν στο δικαστήριο και βεβαίως ε, αμφισβήτησαν ε, τις απόψεις και των δυο μας. Η απόφαση. Η απόφαση είναι πάρα πολύ θετική, όχι μόνο για την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, πρέπει να πάμε παραπέρα και να πούμε ότι είναι θετική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλα τα θεσμικά όργανα, με την έννοια ότι το δικαστήριο θεώρησε ότι ο κύριος όγκος της συμφωνίας στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και για τις υπηρεσίες μεταφορών και το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη που έχει βεβαίως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό επιβεβαιώνει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης ε, στην εμπορική πολιτική μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα μας βοηθήσει, όπως είπατε κι εσείς, στο να ξανασχεδιάσουμε το μέλλον των ε, συμφωνιών ελευθερίου Όπως είπε ήδη η Επίτροπος όταν την ρωτήσατε, τώρα χρειάζεται χρόνος να αναλύσουμε προσεκτικά αυτή την γνωμοδότηση για τη μελλοντική μας πολιτική εμπορίου και επενδύσεων και άρα σήμερα θα σας απογοητεύσω γιατί θα αναφέρω μόνο τα πιο σημαντικά τμήματα αυτής της απόφασης και δεν είμαι έτοιμος σήμερα, ούτε έχω την εντολή ε, να πάω παραπέρα από αυτό τις πιθανές επιλογές δηλαδή, αλλά νομίζω ότι αρκετές ακούστηκαν ήδη και πρέπει να μελετήσουμε τώρα και εντός της Κομισιόν ε, και με εσάς και με τα κράτη-μέλη πριν ε, καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, σύντομα, τι είπε το δικαστήριο ακριβώς να σας ε, πω τα βασικά στοιχεία της γνωμοδότησης. Το δικαστήριο θεωρεί ότι οι εξής διατάξεις είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ε, Ένωσης. Εμπόριο αγαθών και ρυθμιστικά ζητήματα, εμπόριο υπηρεσιών και οι τέσσερις τρόποι, ε, πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιες προμήθειες, ανταγωνισμός, πρόσβαση στην αγορά των επενδύσεων, άμεσες ξένες επενδύσεις, προστασία επενδυτών μόνο στο βαθμό που αφορά άμεσες ξένες επενδύσεις, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη και όλες οι διατάξεις διαφάνειας. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ε, υπό το άρθρο 207 στην κοινή εμπορική πολιτική δηλαδή της συνθήκης και το δικαστήριο αποφάσισε και αυτό νομίζω είναι σαφές και σημαντικό για το μέλλον ότι όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν το εμπόριο καθώς στόχο έχουν να προωθήσουν, να διευκολύνουν ή να καθορίσουν το εμπόριο και έχουν άμεσα αποτελέσματα από το εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι στην παράγραφο 36 της γνωμοδότησης και βασίζεται ακριβώς σε αυτό το δικαστήριο στο να διατρέξει όλα τα κεφάλαια και να καταλήξει τα συμπεράσματα του. Είναι επίσης αξιοσημείωτη η απόφαση αυτή όσον αφορά το κεφάλαιο 13 για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη και τις υπηρεσίες μεταφορών που συζητήθηκε πάρα πολύ ενώπιον του δικαστηρίου και όπου τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο είχαν διαφορετική από... άποψη από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Το δικαστήριο αποφάσισε το κεφάλαιο αυτό περί βιώσιμης ανάπτυξης εμπίπτει στην κοινή εμπορική πολιτική, καθώς η πολιτική αυτή ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συνθήκη, την βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ θετική αυτή η σαφήνεια. Επίσης, συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα των υπηρεσιών μεταφορών όπως αναφέρει και η παραγραφός 5 ε, της ε, σύμβασης η οποία αποκλείει ρητά ε, το πεδίο των μεταφορών από την εμπορική πολιτική. Εδώ πέρα λοιπόν το δικαστήριο βασίστηκε στην λεγόμενη αρχή Χερτά που βασίζεται σε μια απόφαση του 1971 και αποφάσισε ότι λόγω της υφιστάμενης εσωτερικής ε, κοινοτικής νομοθεσίας και εδώ έχει η κοινότητα αποκλειστική αρμοδιότητα. Και με την ομοδότηση αυτή του δικαστηρίου ολοκληρώθηκε μια δύσκολη και οδυνηρή συζήτηση με το Συμβούλιο για τις Υπηρεσίες Μεταφορών. Και αυτό καλύπτει και την προμήθεια τέτοιων υπηρεσιών και βεβαίως κατέληξε παρόμοιο συμπέρασμα για τις διακρατικές ε, επιλύσεις διαφορών. Τώρα, αυτά αφορούσαν την αποκλειστική αρμοδιότητα. Για την αποκοινού αρμοδιότητα. Ενώ επιβεβαίωσε λοιπόν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, για τις έμεσες ξένες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου δηλαδή, και το πιο σημαντικό για το μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών, ε, είπε ότι υπάρχει κοινή αρμοδιότητα ε, σύμφωνα με το άρθρο 207 ε, όπου αναφέρεται, αναφέρονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Άρα οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής αλλά στην ελεύθερη ε, κίνηση κεφαλαίων. Και αυτό είναι κοινή αρμοδιότητα. Η ανάλυση του δικαστηρίου για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών επίσης είναι καινοτόμος και για εμάς και τώρα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα ερμηνεύσουμε αυτά τα ευρήματα. Σε μια ευρύτατη δήλωση που υπάρχει στην παράγραφο 292 της γνωμοδότησης, το δικαστήριο λέει ότι το να φύγουν οι διαφωνίες από τα δικαστήρια των κρατών μελών, κατ' οποίο οποίο κανίστιες, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την συνένεση των κρατών μελών. Μια ξεκάθαρη δήλωση λοιπόν που μας προξενεί έκπληξη εμείς είχαμε διαφορετική άποψη και επίσης και ο Γενικός Αγγελέας είχε διαφορετική άποψη. Και γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο το τι σημαίνει αυτό και τι αντίκτυπο θα έχει στο μελλοντικό σχεδιασμό των συμφωνίων μας. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση. Είναι η πρώτη απόφαση στην οποία το Δικαστήριο ερμηνεύει τις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας για την ε, εμπορική πολιτική και δεν είναι υπερβολικό νομίζω να πούμε ότι πραγματικά αφορά την ουσία της εμπορικής ε, πολιτικής ε, και βέβαια σε μεγάλο βαθμό παρακολούθησε τις απόψεις του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν το Δικαστήριο και έτσι έλυσε ζητήματα τα οποία μας ενοχλούσαν επί σειρά ετών. Πρόκειται λοιπόν για μια ευρύτατη ερμηνεία των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και θεωρεί ότι δεν υπάρχει ε, πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών πια. Κάτι επίσης διαφορετικό από αυτό το οποίο είπε ο Γενικός Εισαγγελέας. Και οι μόνες κοινέ αρμοδιότητες που υπάρχουν είναι το ISDS και οι έμεσες επενδύσεις. Όπως είπα, θα το συζητήσουμε αυτό πρώτα απ' όλα εντατικά εντός της Κομισιόν, κάτι το οποίο νομίζω θα μας πάρει μερικές εβδομάδες και μετά ευχαριστώ, θα επιστρέψουμε ε, για να δούμε τι θα κάνουμε με το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την νομική υπηρεσία της Κομισιόν. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις? Όχι. Μετά θα α, ε, ρωτήσω την δική μας νομική υπηρεσία. Έχει παρατηρήσεις? Όχι. Η οποία έκπληξη. Παρακαλώ. Αν θέλετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αλλά η Κομισιόν είπε τα ουσιώδη. Το μόνο που θα τονίσω είναι ότι υπήρχαν κάνα δύο θέματα που υπήρχε έντονη άποψη των κρατών μελών και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είχαν διαφορετική άποψη για τις μεταφορές που αποκλείονται. Αλλά για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται εδώ υπάρχουν κοινοί κανόνες που μπορούν να επηρεαστούν. Επομένως, εντάσσονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα. Γενικά θα περιμέναμε να είναι ε, οι δεσμεύσει που έχουμε και σε άλλε συμφωνίε. Αλλά θα πρέπει να το δούμε ίσω ε, και στι μελλοντικέ ε, συγκεκριμένε συμφωνίε που αφορούν αυτού του συγκεκριμένου κοινού κανόνε. Πολύ σύντομα επίση, η βιώσιμη ανάπτυξη. Αντίστοιχα, τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο είχαν τελείω διαφορετική άποψη από εμά. Αυτέ οι δεσμεύσει επιβεβαιώνουν τι δεσμεύσει που έχουν αναλυθεί ήδη σε διεθνεί συμφωνίε. Και ακριβώ για αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο θεώρησαν ότι θα ήταν εθνικές αρμοδιότητες. Όμως το δικαστήριο δεν το δέχτηκε αυτό. Δεν δέχτηκε αυτό το επιχείρημα. Καλύτερα να βάλω εδώ μια τελεία. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής έχει τώρα το λόγο για την Σιγκαπούρη. David Martin, σύντομο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Βλέπετε αυτή τη στιγμή πως το Brexit αλλάζει την προπτική που έχουμε για διάφορες συμφωνίες. Ξέρετε ότι η απόφαση αυτή φάνηκε σε πάρα πολλά πρωτοσέλιδα του Βρετανικού τύπου, ιδίως σε αυτούς οι οποίοι είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και ελέγχθη ότι ε, η απόφαση αυτή ουσιαστικά θα διευκόλυνε μια μελλοντική εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του Ηνωμένου Βασιλείου. Βέβαια η οπτική γωνία διαφοροποιείται πάρα πολύ από το που βρίσκεται κανείς. Ακούσαμε την Επίτροπο. Εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά η απόφαση αυτή του δικαστηρίου πραγματικά μπορεί να μας σώσει από κάποια προβληματικά σημεία που υπάρχουν στα πλαίσια της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η απόφαση αυτή και να μπορέσουμε στο μέλλον για κάποιες συμφωνίες να διαχωρίζουμε το εμπορικό κομμάτι από το επενδυτικό το κομμάτι. Υπάρχουν έπειτα και τα κεφάλαια εκείνα που έχουν να κάνουν με την βιώσιμη ανάπτυξη, για τα οποία το δικαστήριο είπε ότι αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα τη εμπορική συμφωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική δήλωση και για τι μελλοντικέ συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τώρα τη Σιγκαπούρη. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή πλέον έχουμε την απόφαση αυτού του δικαστηρίου, θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε γρήγορα με την απόφαση αυτή. Ξέρετε ότι περίμενε η πλευρά της Σιγκαπούρης τρία επιπλέον χρόνια μόνο και μόνο για να εκδοθεί αυτή η απόφαση από το δικαστήριο και αυτό λόγω εσωτερικών προβλημάτων πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα και προκειμένου να γίνει αυτό, το λέω για τρίτη φορά, πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο αυτά τμήματα, εμπορικό και επενδυτικό τμήμα. Και όσον αφορά το ιστορικό που έχουμε με τις επενδυτικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη, 47 επενδυτικές συμφωνίες με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμία χώρα ουσιαστικά δεν εστράφει ποτέ κατά της Σιγκαπούρης, ουδέποτε έγινε κάποια προσφυγή, ενώ η, προσφυγή, η είχε κάνει δύο προσφυγές κατά της Ινδονησίας και μία κατά του Μιανμάρ. Νομίζω λοιπόν ότι ε, και αυτό καταδεικνύει ότι θα πρέπει να έχουμε το στομότερο δυνατό μια εμπορική συμφωνία με την ε, Σιγκαπούρη. Ενδεχομένω, όπω σα είπα, διαχωρίζοντα το εμπορικό από το παιδιτικό κομμάτι. Ενδεχομένω να προχωρήσουμε μόνο με την εμπορική συμφωνία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιο, ενδεχομένω αν υπάρχει και κάποιο εδώ πέρα από την πρεσβεία τη Σιγκαπούρη, να πει επίσημα προ την ε, πλευρά τη Σιγκαπούρη ότι σε ευχαριστούμε για την υπομονή του. Πρόεδρος, η ε, ευρωπαϊκή πλευρά είναι αυτή που έθεσε το κεφάλαιο αυτό το επενδυτικό, δεν ήταν ε, η πλευρά της Σιγκαπούρης. Πολύ ωραία. Μπορούμε να ακούσουμε τώρα πρώτα τους συντονιστές και συνέχεια άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Δύο λεπτά ο καθένας και ξεκινάμε με τον κύριο Κάσπερη. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς ως ΕΛΚ είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη που ε, μας έδωσε το ΔΕΚ και είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται πιο δημοκρατική όταν το κάθε φόρουμ αποφασίζει για τα πάντα. Όπως ακριβώς ε, όταν ένα δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του χωρίς να μας ρωτήσει, νομίζω και εμείς είμαστε δημοκρατικοί όταν λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς να ρωτάμε τα άλλα επίπεδα. Δεύτερον, θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι θα κάνουμε προσεχώς με το θέμα των επενδύσεων. Θέλουμε όντως μία ξεχωριστή συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων ή θέλουμε μία συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων που δεν θα έχει επίλυση διαφορών και θα κάνουμε μια έξτρα συμφωνία που πρέπει να κυρωθεί από τα κράτη-μέλη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον να το σκεφτούμε. Και δεύτερον, μου έκανε εντύπωση η διατύπωση του προσώπου της Κομισιόν ε, για τα δικαστήρια επίλυσης ε, εμπορικών διαφορών είπε ε, την λέξη removing ότι αφαιρούνται αρμοδιότητες από τα εθνικά δικαστήρια. Πρέπει εδώ πέρα νομίζω να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βρούμε κάποιες δημιουργικές λύσεις για το πώς θα υπάρχει δυνατότητα να προσφεύγουμε στα δικαστήρια για την προστασία των επενδύσεων και βεβαίως ε, την προσφυγή σε ένδικα μέσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν ακριβώς να συζητήσουμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα τις ε, επόμενες εβδομάδες. Αλλά α, ε, χαίρομαι που 8 χρόνια μετά τη θέση ενισχύει τη συνθήκη της Λισαβόνας επιτέλους ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητές μας. Ευχαριστώ. David Martin τώρα. Ε, ευχαριστώ εκπρόσωπο του συνάδελφο το ένα θέμα το οποίο δεν ανέφερα που θα ήθελε να τονίσει. Καλωσορίζω οπωσδήποτε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά ε, δεν θα πρέπει να ε, θεωρούν τα κράτη-μέλη εκεί όπου έχουν μεικτή αρμοδιότητα ότι μπορούν να κάνουν διμερείς ε, συμφωνίες ούτε για το ενεργειακό κεφάλαιο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές είναι τοξικές ιδέες, πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ε, μεταρρύθμισης. Νομίζω το δέχτηκε ούτως ή άλλως η Επίτροπος. Για εμάς η επιτροπος για εμας μεταρρυθμιση των επενδυτικών ε, συμφωνιών ε, δεν έχει τελειώσει. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι οι επενδύσεις πρέπει να είναι μια ξεχωριστή αρμοδιότητα. Σας ευχαριστώ κύριο Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι πολλοί από εμάς ε, εξεπλάγησαν από την απόφαση. Ήταν ε, ενδιαφέρουσα, βέβαια, κυρίως γιατί δεν ακολουθήθηκε η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα. Αλλά βεβαίως ε, τα πράγματι, όπως είπαν οι συνάδελφοι, τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες σοβαρές ερωτήσεις. Να επανέλθω εγώ σε κάτι. Εγώ ήμουν εισηγητής για αυτό το θέμα μέχρι το 2014 και ελπίζαμε τότε μέχρι το 2014 να έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία και η Σιγκαπούρη ήταν πολύ υπομονετική, δεν τους φερθήκαμε σωστά. Δηλαδή ε, νομίζουν και οι δύο πλευρές ότι έχουν υπογράψει μια συμφωνία και μετά πάμε και την ξανανοίγουμε και λέμε «Α, συγγνώμη, τι να κάνουμε τώρα, άμα θέλετε». Ήταν άδικο, νομίζω και οι Σιγκαπούροι μας φέρθηκαν πολύ εντάξει και θα πρέπει να τελειώσουμε τη συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Και το επόμενο θέμα, αν περιλαμβάνει έναν ξεχωριστό μηχανισμό επίλυση διαφόρων για να τελειώσουμε με αυτή τη συμφωνία, πρέπει να το κάνουμε και η ομάδα μου δεν έχει ακόμα θέση για το αν θα πρέπει να γίνεται χωριστό αυτό για κάθε συμφωνία, αλλά ε, ίσως θα πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση, γιατί κάποιες χώρες σαφώς ε, δεν αποτελούν ζήτημα για τις επενδύσει και μπορούμε να τι εμπιστευτούμε. Για άλλες χώρε. Ε, για κάποιες χώρες, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν χρειάζεται αυτό το κεφάλαιο. Γιατί έχουν το σωστό νομικό πλαίσιο, αμοιβέ, αρμοδιότητα κτλ. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση. Αλλά γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί ε, θέλουν ακριβώς να ακολουθούν κάποια υποδείγματα συμβάσεων. Και ακριβώς για τον μηχανισμό ε, επίλυση διαφορών θέλουν οι Αμερικανοί να ακολουθήσουμε το ISPS. Είναι λοιπόν ε, σημαντική αυτή η συζήτηση, όχι μόνο εδώ, αλλά παγκοσμίω. Hopefully... Σύντομα, γιατί ο Ραμόν έρχεται όπου να είναι ε, και εκπροσωπεί την ομάδα μας για το θέμα τη Συγκαπούρη. Καλή είναι η σαφήνεια πάντα, ο σεβασμός των κανόνων και η σαφήνεια των κανόνων είναι πολύ σημαντικό πράγμα και σε ό,τι αφορά το εμπόριο ελπίζω όλοι να δεχτούν τις ε, νομικές πτυχές και να μην ε, ασκήσουν μικροπολιτική με όπλα αυτές. Υπάρχουν όμως πολλά πολιτικά θέματα ανοιχτά. Το δικαστήριο δεν απάντησε τις πολιτικές ερωτήσεις και δεν είναι και ρόλος να το κάνει. Νομίζω ότι απόκειται το Συμβούλιο τώρα πρωτίστως να αξιολογήσει τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τις μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίες. Ε, να δώσει σαφείς εντολές Φερρυπίν, να εμπλέκει τα Εθνικά Κοινοβούλια Φερρυπίν. Ε, να εμπλέκονται οι πολίτες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας πιο ενεργά κτλ. Γιατί μερικές φορές λέγεται και σε συζητήσει εδώ στο δικαστήριο ότι θα πρέπει το δικαστήριο να ξεκαθαρίσει ποιος έχει λόγο στις εμπορικές πολιτικές πότε και σε ποιες περιπτώσεις. Ποτέ όμως δεν πρέπει να είναι. Δεν γίνεται αυτό και δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η πολιτική ηγεσία τώρα, να, τα πολιτικά θέματα να ξεκαθαριστούν, ούτως ώστε να μπορέσει να εργαστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με σεβασμό του, πνευμα, του πνεύματος της Λισαβόνας, ε, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή που έχουμε πάρα πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τους κανόνες για το εμπόριο, ε, για ένα εμπόριο δηλαδή που να βασίζεται σε κανόνες, αλλά και για να αρπάξουμε και τις ευκαιρίες. Πρέπει όμως ε, αυτές τις ευκαιρίες να τις ε, εκμεταλλευτούμε μόνο εάν υπάρχει πολιτική ας πούμε, βούληση. Τώρα, μια και ξεκαθαρίσαμε τα νομικά, ας δούμε τώρα τι γίνεται και με, την, ε, με τα πολιτικά θέματα για την επόμενη φάση. Από την ΚΟΕ, η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα ήθελα να αναφέρω για την σύμβαση αυτή. Το πρώτο είναι ότι οι συμβάσεις με επιδιαιτησία πρέπει να υποβληθούν στα κράτη-μέλη και αναφέρω εδώ πέρα την παράγραφο 292 γιατί διαφέρουν ε, από τις νομικές αρμοδιότητες των κρατών μέλων. Και θα πρέπει, όπως ε, λέει εδώ πέρα, ότι αφαιρούνται αρμοδιότητες από τα δικαστήρια των κρατών μελών. Ελπίζω λοιπόν να μην συμβεί αυτό. Δεύτερον, το δικαστήριο είπε ερητός ότι δεν εξετάζει το εάν είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτή η διαδικασία επίλυσης διαφορών. Δεν είναι ακόμα σαφές και πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία στο πρωτοβουλίο της Βαλωνίας και θα δούμε τι θα γίνει και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Τρίτον, δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο να ε, μην μπορούν να υποβάλλονται στις εθνικές κυβερνήσεις οι συμβάσεις για πολιτικούς λόγους. Το είδαμε και με την ΣΕΤΑ και το ISDS οπωσδήποτε. Εμείς ε, πέρα από αυτό βλέπουμε και άλλα προβλήματα. Παραδείγματο χάρη η regulatory cooperation και οι διαφάνειες διαπραγματεύσεις. Και θα ήθελα επίσης να αντιδράσω στην παρατήρηση του κυρίου Φιέλνερ. Την στιγμή που ε, είναι αντικειμενική παρατήρηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μακριά από τους ε, πολίτες, ότι έχει χαμηλή συμμετοχή στις ε, εκλογές. Ακούμε ότι πρέπει να φύγουν και άλλες αρμοδιότητες από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ο κύριος Χέλνερ απλά αποδεικνύει αυτό το οποίο θέλω να πω. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να φροντίσουμε αν αφαιρεθούν αρμοδιότητες κύρωσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια να ασκήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο και να δούμε βεβαίω και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί αυτό βλάπτει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πρέπει να κλείσει κάποια στιγμή αυτή η ψαλίδα μεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ κύριε Χάτολα για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η αποσαφήνιση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όπως ακούσαμε και βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κινούμεθα όλο και περισσότερο προς εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει από την απόφαση αυτού του δικαστηρίου. Και πιστεύω επίσης ότι ε, τη στιγμή εκείνη που τα κράτη-μέλη ή τα κοινοβούλια τους θα πρέπει να έχουν κάποιο λόγο είναι ότι διαπραγματεύεται η δική τους η έντολη. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα συμπέρασμα της απόφασης αυτής του δικαστηρίου. Αν πραγματικά τα κράτη-μέλη θέλουν να μπορούν να διατηρούν το δημοκρατικό αυτό έλεγχο, πέρα από τον έλεγχο που γίνεται βέβαια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε όταν θα εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές τους εντολές, τότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάποιο λόγο. Και θυμάμαι αυτό το οποίο ζήτησε από την Επιτροπή μας η Επίτροπος Μάλστρομ, ότι εμείς πρέπει αυτή να υποστηρίξουμε στην προσπάθειά της να κάνει τις διπραγματικές αυτές εντολές δημόσια διαθέσιμες, πράγμα το οποίο δεν το ήθελε ποτέ, ξέρετε, το Συμβούλιο. Τότε λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνουν δράση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει πλέον μια σαφήνεια όσον αφορά την φύση των κεφαλαίων αυτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό διότι θα δώσει περισσότερες ε, δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθήσει περισσότερο την εταιρική ευθύνη σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί πολύ συχνά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη διστάζουν πάρα πολύ να πάρουν αυτό το δρόμο, να κινηθούν προς αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φεγόν τώρα για το INF. Αγαπητοί συνάδελφοι, θαύμα έλαβε χώρα από ό,τι βλέπω. Και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε μια πολύ σημαντική προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αναφέρθηκε σε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας όμως ότι κάθε συμφωνία έχει ένα χαρακτήρα μεικτό ή ένα χαρακτήρα με συντρέχουσες αρμοδιότητες και στη συνέχεια θα πρέπει να αποφαίνονται και τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω λοιπόν ότι επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο εξ αρχής θέλαμε, όσον αφορά δηλαδή τη δυνατότητα ελέγχου. Και όσον αφορά τη Συμφωνία της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο να αποσύρουμε από, να αποσύρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, αποκλειστική εντολή διαπραγματεύση διαπραγμάτευσης που έχει, η οποία μας έφερε στην πολύ αυτή δύσκολη θέση, σε αυτό το αδιέξοδο. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούν τα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια να διαπραγματεύεται βάσει των πραγματικών συμφερών της Ένωσης και όχι βάσει των συμφερών των ομάδων πίεσης. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την απόφαση αυτού του δικαστηρίου, συζητητής για το ζήτημα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε κολλήσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε καμία πρόοδος, το είπαν αυτό πολλοί συνάδελφοι και τώρα βλέπω ότι θα καταφέρουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να εγκρίνουμε τελικά τη συμφωνία αυτή το συντομότερο δυνατό. Λοιπόν, πώς έγινε δεκτή η απόφαση αυτή στη Σιγκαπούρη καταρχάς, αυτό πρέπει να δούμε και πώς θα μπορέσει εν συνεχεία να εφαρμοστεί. Δεύτερον, Νομίζω ότι αναφερόμενο στους δύο τελευταίους ομιλητές θα πρέπει να πω το ακόλουθο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την αποκλειστική αρμοδιότητα που ούτως ή άλλως είχε, η οποία πιστεύω ότι έχει ενδυναμωθεί αυτή τη στιγμή με την απόφαση του δικαστηρίου και μπορεί πραγματικά να αναλάβει πλήρως ευθύνες, ίσως όχι μόνο σε σχέση με τη Σιγκαπούρη, αλλά και σε σχέση με τη συμφωνία που θα συνάψει με άλλες χώρες. Και τέλος, να θέσω ένα ερώτημα. Στα πλαίσια του ISDS, της επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, θα μπορούσαμε να είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πολυμερές επίπεδο, να έχουμε δηλαδή ένα υπόδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διεθνώς και το οποίο στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε και για τις επόμενες συμφωνίες, τις μελλοντικές συμφωνίες. Γιατί Όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για έλλειψη διαφάνεια και επιστροφή στα εθνικά κοινοβούλια πιστεύω ότι θα κάνουν κάθε το δυνατό για να παρεμποδίσουν αυτέ τι συμφωνίε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το δικαστήριο μα δίνει πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα και να προωθήσουμε περισσότερε τέτοιε συμφωνίε. Ο κύριο Φιένερ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που και ο κύριο Καμάλο αναφορά την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι στα πλαίσια των διαπραγματευτικών εντολών που έχουμε για συμφωνίες δεν έχω ξαναδεί τέτοιες εξελίξεις. ξεκινήσαμε όντως με μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, στη συνέχεια είπαμε «Α, η συνθήκη της Λισαβόνα θέλει να περιλαμβάνουμε τώρα και τις επενδύσεις». Κάνουμε και την επενδυτική συμφωνία, σφίξαμε χέρια, βάλουμε υπογραφές και μετά πάμε στην Καπούρη και τους λέμε «Ξέρετε, αλλάξαμε τώρα γνώμη, ας αλήξουμε πάλι την συμφωνία εξ αρχής». Και σαν να μην έφτανε αυτό, η σοφία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι θα έπρεπε επί της ε, συμφωνίας αυτής, τη συγκεκριμένη με τη Σιγκαπούρη, να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Ενώ για τον Καναδά είπαμε ότι θα έπρεπε να αποφασίσει το Συμβούλιο. Με αποτέλεσμα τελικά να εφαρμοστεί πολύ πιο γρήγορα συμφωνία με τον Καναδά και ακόμα νεκρεμεί, ακόμα νεκρεμεί μετά από τόσο καιρό η συμφωνία αυτή με τη Σιγκαπούρη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν να στήσουμε συγγνώμη τη Σιγκαπούρη. Δεύτερον, να υποσχεθούμε ότι ουδέποτε θα κάνουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Δεν δικαιούμεθα να κάνουμε κάτι τέτοιο μόνο και μόνο επειδή είναι μια μικρή χώρα, μια μικρή αν θέλετε συμφωνία. Στα πλαίσια τη συμφωνία αυτή με τη Σιγκαπούρη, προφανώ θα πρέπει να δούμε πώ εξελίχθουν τα πράγματα στο μέλλον και πώ η συμφωνία αυτή θα επηρεάσει μελλοντικέ συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ακούσουμε όμω και το δικαστήριο, να προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με του κανόνε και να εγκρίνουμε μελλοντικέ διαπραγματευτικέ εντολέ κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολείται αυτή ω πλέον αρμόδια με την εμπορική πολιτική τη. Ένα ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Τι κάνουμε με τι υφιστάμενε, τι τρέχουσε εντολέ. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να είχαμε δύο διαφορετικέ συμφωνίε βάσει τη ίδια εντολή. Από πρακτική δηλαδή πλευρά, πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι δυνατότητε που μα δίνονται. Θα κλείσω τον κατάλογο μιλητών. Έχουμε πέντε ακόμα άτομα. Κάρολ. Ευχαριστώ. Ήθελα να επανέλθω η λέξη που αναφέρθηκε σήμερα περισσότερο ήταν η σαφήνεια. Πράγματι ξεκαθάρισαν οι αρμοδιότητες, αλλά θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει νομίζω και το εάν το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν έγινε σε αυτήν την διαδικασία. Ίνμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Φέρνερ μόλις τώρα. Ότι στην περίπτωση της Σιγκαπούρης θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με τον Καναδά. Να κάνουμε δηλαδή μία επικύρωση και να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή η συμφωνία και μετά να επικυρώσουν τα κράτη-μέλη των υστέρων για να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία της συμφωνίας με τη Σιγκαπούρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνεται με τη Σιγκαπούρη αυτό που γίνεται με τον Καναδά. Ε, η βασική ερώτηση όμως είναι τι κάνουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η απόφαση διευκρινίζει την, τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ περι, περισσότερες περιπτώσεις από αυτές που είχε προτείνει ο Γενικός Εγγελίας αρκετά αρχικά. Και για το εμπορικά θέματα και για, τα, για τις επενδύσεις ε, χαρτοφυλακίου και τις επενδύσεις ε, κρατών. Όλα αυτά διευκρίνησε. Εμείς θα ήθελα να αναλύσουμε τα υπέρ και τα κατά κάθε διαδικασία που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και σε ποιο βαθμό μπορούμε τις επενδύσεις να τις χωρίσουμε εντελώς από το εμπορικό κεφάλαιο ε, στις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολυμέρεια στο, στα επενδυτικά δικαστήρια. Για να λειτουργούν με ένα πολυμερή τρόπο και να μπορούν να επιλύουν οποιαδήποτε σύγκρουση, ε, οποιοδήποτε επενδυτή. Οποιοδήποτε και αν το μοντέλο που θα επιλέξουμε. Δεν ξέρω αν έχει νόημα ίσως να ζητήσει το Κοινοβούλιο να γίνει μια μελέτη για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κ. Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρα από, τα, από τις επιπτώσεις που έχει η απόφαση, το, τη στιγμή που θα καθορίσουμε τη φύση των συμφωνιών, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα ε, που έθεσα και στην Επίτροπο, ε, στο θέμα του χρονισμού. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι, με, αυτό το, με αυτή τη διαδικασία είναι σχεδόν αδιανόητες. Ε, δηλαδή θέλουμε καταρχάς την διαπραγματευτική εντολή ένα με τρία χρόνια. Μετά θέλουμε έγκριση για διαπραγμάτευση και να, διαπραγματεύσεις που φτάνουν και τα 20 χρόνια. Για τα μερικοσούν έχουμε τελειώσει ακόμα. Και μετά μια επικύρωση ε, που στα κράτη-μέλη θέλουν, θέλουμε δύο χρόνια. Εμείς τα κάνουμε πιο γρήγορα. Έτσι. Και αν μετά γίνει και προσφυγή στην ε, δικαιοσύνη, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα στο άπειρο, ας πούμε. Αενάω να ασχολούμαστε. Δεν είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στου συνομιλητέ μα, όπω δεν είμαστε αξιόπιστοι αυτή τη στιγμή απέναντι στο Μερκοσούρ. Και χάνουμε και διάφορε ευκαιρίε. Η Επίτροπο ανέφερε, απαντώντα το ερώτημα που έθεσα εγώ, το θέμα ότι, είναι, ότι γίνονται πλέον ε, άχρηστες αυτές οι συμφωνίες. Μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, λογικό είναι να κάνουμε μία συζήτηση για τις, α, τις προθεσίες. Γιατί αν μπερδευτούμε μέσα στις, στους δεδάλους των δικών μας των διαδικασιών, χάσαμε. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα στοιχείο εξορθολογισμού εκεί μέσα. Ε, το είπε και η Επίτροπος. Εμείς δεν είμαστε ο πιο αργός κρίκος αλυσίδας, αλλά πρέπει συνολικά να κάνουμε όλη μια προσπάθεια τόσο ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία η οποία μας κάνει να χάνουμε πολύ από την αξιοπιστία μας απέναντι στους ε, συνομιλητές μας. Ο κύριος Τρεμόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που ήρθα αργά γιατί καθυστέρησα στην Επιτροπή για το, τα θέματα με τον Παναμά. Το Παναμά Ήθελα να μιλήσω για τα θέματα που αφορούν ε, τη Σιγκαπούρη. Συμφωνώ με τον κύριο Σαλαφράγκα μετά όσα είπε στο τέλο. Εγώ ήθελα μια, πάντα μια γρήγορη επικύρωση των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Καταρχά, γιατί όλοι κερδίζουν. Κερδίζουν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, όλοι εξάγουμε στη Σιγκαπούρη. Επομένω, ε, ήταν ξεκάθαρη υπόθεση αυτή. Που θα μπορούσαμε να την πουλήσουμε στου πολίτε, να εξηγήσουμε στου πολίτε μα γιατί χρησιμεύε. Και τώρα χρειαζόμαστε επικύρωση από τα κράτη-μέλη, χάνουμε και άλλο χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σαλαφράκα, λοιπόν, που ότι χρειάζεται να γίνεται μία συζήτηση για το πώ θα επιταχύνουμε τη διαδικασία για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία που χάνουμε. Γιατί εκπροσωπούμε και του πολίτε εδώ πέρα. Και θα πρέπει, αν τώρα θα πρέπει να δώσουμε φωνή και στα κράτη-μέλη, τότε εμεί ποια προστιθέμενη αξία φέρνουμε εδώ πέρα. Μια και εμεί μπορούμε να επιταχύνουμε. Εμεί οι ίδιοι διαπραγματευόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Τι νόημα έχουμε εμεί τότε. Πρέπει να διαρωτηθούμε τι συμβαίνει εδώ. Και φυσικά, αν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, σε αυτή την περίπτωση εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση τα κράτη-μέλη να έχουν το τελευταίο λόγο. Ο κύριο Σόλτ. Uh, Ευχαριστώ, Μπέρντ. Νομίζω αυτό απευθύνεται στο Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο διαμορφώνει την εμπορική πολιτική και εδώ νομίζω πως η απόφαση μας δίνει ένα πολύ καλό επιχείρημα, ότι πρέπει οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων πριν τεθούν ενισχύ, πρέπει να συζητηθούν στα κράτη-μέλη το πώς δηλαδή οι υπουργοί διαμορφώνουν μια εντολή πρέπει να επανέλθει, να επανασυνδεθεί με τα κοινοβούλια και την κοινή γνώμη των χωρών. Και εδώ πέρα συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Χάουταλα. Εδώ πρέπει να ξανασκεφτούμε το πώς θα οργανώσουμε την εμπορική πολιτική. Τώρα δεν είναι δικιά μας η δυνατότητα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι αντίκτυπο έχει η εμπορική πολιτική στην πραγματική ζωή στα κράτη-μέλη. Και τότε μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις και πώς θα εφαρμόσουμε τα αποτελέσματά τους υπό μορφή συνθήκης, συμφωνίας κτλ. Είτε είναι η συμφωνία αγαθών είτε επενδύσεων. Και στις δύο περιπτώσεις νομίζω έχουμε ευθύνη να δίνουμε αναφορά, αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι κάνουμε ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έχουμε μια ξεκάθαρη ευθύνη νομίζω μετά από την απόφαση του δικαστηρίου και ελπίζω με το αποτέλεσμα αυτό να κωδικοποιήσουμε την εμπορική πολιτική όπως είπε η κυρία Ρέντινγκ στην Επίτροπο, δηλαδή ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο κατά το οποίο σημαίνει, σημαίνει να λάβουμε υπόψη τις απόψεις των πολιτών και τις επιθυμίες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να σκεφτούμε πράγματι το τι θα γίνει με αυτή την απόφαση. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης το επενδυτικό δικαστήριο. Γιατί είναι σαφές ε, πως οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Ε, αυτό φαίνεται από το άρθρο 207, αλλά τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που λέει ότι το δικαστήριο αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης γιατί αφαιρείται αφαιρεί αρμοδιότητες από τα εθνικά δικαστήρια ε, θα μπορούσαμε σε αυτό να αντιπροτείνουμε ότι μπορεί κάτι να πάει σε αυτό το επίπεδο όταν εξαντληθεί εξαντληθούν τα εθνικά ένδικα μέσα. Και ο κύριος Κασφάρη επίσης έκανε κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πολλές ερωτήσεις λοιπόν. Θέλει η Κομισιό να απαντήσει κάποιες από αυτές. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε. Να μιλήσω τώρα αγγλικά. Πολλές ερωτήσεις πακούστηκαν, ακούστηκαν, θεμητές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω ομαδοποιώντας τες. Οι πρώτε είχαν να κάνουν με τη Σιγκαπούρη. Τι θα γίνει με τη Σιγκαπούρη. Προφανώς είμαστε σε επαφή με την πλευρά της Σιγκαπούρης. Τους εξηγήσαμε το υπόβαθρο της, συζήτη, της απόφασης αυτής του δικαστηρίου. Εξηγήσαμε για ποιο λόγο είχαμε την καθυστέρηση αυτή, για ποιο λόγο επελέξαμε αυτή τη συμφωνία, επειδή ήταν η πρώτη, η πρώτη η οποία υποβλήθηκε στο Συμβούλιο προς έγκριση μετά την θέση ενισχύ της της Αβώνας. Ήταν η πρώτη τέτοια συμφωνία. Δεν μπορούσαμε λοιπόν εμείς να παρακάμψουμε, αν θέλετε, τη συμφωνία αυτή, γιατί ουσιαστικά δεν θα καταφέρναμε τελικά να ερμηνεύσουμε σωστά τη συνθήκη. Και η πλευρά της Σιγκαπούρης είχε ζητήσει να υπάρχει ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο που έκανε με τις επενδύσεις. Δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία επενδύσεις, ήταν αρχική πρωτοβουλία της Σιγκαπούρης. Και βέβαια δεν υποφέρει μόνο η Σιγκαπούρη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την καθυστέρηση αυτή. Καταλαβαίνω ότι είναι πόδινο αυτό για όλους, αλλά αν δείτε τι κερδίζουμε τελικά μέσω της ε, καθυστέρησης αυτής, θα συνειδητοποιήσετε τελικά ότι είναι μια επένδυση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, η οποία είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές. Ο πρόεδρο Επιτροπή Μπαρόσο τότε ήταν αυτό ο οποίο αποφάσισε να προσφύγει στο δικαστήριο για την ερμηνεία. Και τελικά η ερμηνεία αυτή είναι θετική και για τι δύο πλευρέ για πάρα πολλέ πτυχέ. Έχω σημειώσει παρατηρήσεις και τι ερωτήσει σας, θα τις αναλύσουμε περισσότερο. Να πω εν συντομία κάποια πράγματα όσον αφορά την πολυπλοκότητα της συμφωνίας αυτής. Είπατε ότι οποιαδήποτε διαιτησία αποκλείεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο οι διακρατικές διαδικασίες αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, δε το δικαστήριο. Λέει επίσης ότι για την προστασία της άμεσης ξένης επενδύσης, την πρόσβαση στην αγορά και αυτά αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το επενδυτικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και μόνο οι διατάξεις εκείνες που έχουν να κάνουν με την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους. Και αν ξέρετε, αυτές είχαν εξαγριώσει, με συγχωρείτε, ορισμένους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με όλες τις επενδύσεις και όλες τις πτυχές των επενδύσεων. Και θα έλεγα ότι το πιο ευαίσθητο ζήτημα είναι η πολιτική διάσταση της συζήτησης αυτής και θα ήθελα εδώ πέρα να συμφωνήσω με αυτά που είπαν η κυρία Χάουτα αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Εν τέλει, τελικά η συζήτηση αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση. Και έτσι ξεκίνησε κιόλα. Υπάρχουν πολλοί που επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βρήκε διάφορα νομικά τεχνάσματα για να αποφύγει τη δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει όμω αυτό με κάποια πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει να κάνει με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει εντολών που προέρχονται από το Συμβούλιο και περνούν από το δικό σα τον έλεγχο. Νομίζω λοιπόν ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν τελικά το πώς πληρούμε τις υποσχέσεις που δίνουμε προς τρίτες χώρες. Και όταν λαμβάνουμε υποχρεώσεις πρέπει να εφαρμόσουμε, να τηρούμε τις υποχρεώσεις αυτές στη συνέχεια. Η διάσταση δημοκρατική επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, αυτό, είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο στο έγγραφό μας για την παγκοσμιοποίηση αναφερόμαστε στην απόφαση αυτού του δικαστηρίου λέγοντας ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εμείς ε, προφανώς λέμε ότι θα πρέπει να εγγυόμαστε πλήρως την δημοκρατία και αυτό γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε υπόλογοι σε εσάς αποφασίζετε εσείς μαζί με το Συμβούλιο για τις συμφωνίες αυτές, αλλά συμφωνώ και με αυτού που είπαν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να λαμβάνουν πιο προδραστική στάση στο πλαίσιο των Εθνικών Κοινοβουλίων πολύ νωρίτερα, δημοσιεύοντα δηλαδή τι διαπραγματευτικέ εντολέ. Ανέκαθεν το έλεγε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ δεν έχει συμμορφωθεί με αυτό το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή όμω υποβληθούν οι εντολέ και ξεκινήσει μια συζήτηση. Αυτή θα πρέπει να γίνεται καταρχά στα εθνικά κοινοβούλια από πολύ νωρί. Δεν θα πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθεί η συμφωνία, να ολοκληρωθεί η εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε να αρχίσετε να επικρίνετε τη συμφωνία αυτή λέγοντα ότι τα πάντα έγιναν και κλεισμένων των θυρών. Όχι, όλα γίνονται και θα πρέπει να γίνονται με τρόπο εντελώ διαφανή και συμφωνώ με όσους είπαν ότι φέρουμε τεράστια ευθύνη και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη για τον τρόπο με τον οποίο τα επιμέρους κράτη-μέλη οργανώνονται στο προκαταρκτικό αυτό στάδιο της επεξεργασίας των συμφωνιών. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θα πρέπει να περάσει περισσότερο προς τα έξω. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία έθιξαν οι ευρωβουλευτές. Ολοκληρώνοντας να κάνω και ένα θετικό σχόλιο, το ζήτημα των αρμοδιοτήτων στις εξωτερικές σχέσεις είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό και ουσιαστικά πολλές φορές έχει πειράσει αρνητικά τις όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο Συμβούλιο για τις εμπορικές συμφωνίες. Χαίρομαι λοιπόν που έρχεται αυτή η απόφαση του δικαστηρίου για να αποσαφηνίσει τα πράγματα. Δεν επιλύει τα πράγματα από πολιτικής πλευράς, αλλά μας δίνει μια νέα βάση, προκειμένου να μπορούμε τώρα να μιλήσουμε πραγματικά για τα πολιτικά ζητήματα, τα οποία πολλές φορές κρύβονται πίσω από νομοτεχνικά, νομοτεχνικές προσεγγίσεις και παρατηρήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Φιένα. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Σας ρώτησα αν θα μπορούσαμε να είχαμε βάσει μιας και εντολής δύο διαφορετικές συμφωνίες πρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εστώ συγγνώμη, δεν απάντησα σε αυτό. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η διαπραγματευτική εντολή σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει την έκδοση διαπραγματεύσεων. Εμεί πιστεύουμε ότι ακόμα και μια εντολή που δεν αποσαφηνίζει το είδο, ή τον αριθμό των συμφωνιών, εμείς μπορούμε να καταλήξουμε σε διαφορετικές συμφωνίες. Τώρα, από πολιτική πλευράς τα πράγματα περιπλέκονται κάπω. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε μία επαναδιατύπωση των νέων διαπραγματευτικών εντολών για τη Χιλή και για τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, Προσπαθούμε δηλαδή από τώρα να δούμε πώ ήδη στα πλαίσια τη εντολή μπορούμε να δώσουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιε ενδείξει για τη συμφωνία την οποία θέλουμε να πετύχουμε. Για να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο και για να επιβεβαιώσουμε τελικά ότι τα πράγματα όντω έχουν αλλάξει μετά την απόφαση αυτού του δικαστηρίου. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Ενδεχομένω να μην απαντήθηκαν όλε οι ερωτήσει αλλά νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν μια κάποια σύγκληση πλέον απόψεων για το ζήτημα αυτό και αύριο στο γεύμα που θα γίνει για το TPC με τα κράτη-μέλη περιμένω πραγματικά να δω ποια θα είναι η άποψη των επιμέρους κρατών μελών για την απόφαση αυτή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό, αυτό το θέμα συζήτησης, να πω επίσης τμήμα ότι στις 19 Ιουνίου θα έχουμε μια παρουσίαση μια μελέτης για την επενδυτική πολιτική και θα γίνει και μια σχετική συζήτηση για την επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα είναι μια ευκαιρία για να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που ξεκινήσαμε τώρα, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την επενδυτική πολιτική μας μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 5, ψηφοφορία. Ή ε, όχι, 5 και 20, στην ώρα μας είμαστε. 17.20 Λοιπόν, 5 και 20, 5 και 20. Οπότε ξεκινάει η ψηφοφορία. Δεν ξέρω γιατί θορυβείτε. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε σε κάποιες περιπτώσεις ηλεκτρονικά. Γι' αυτό πρέπει να δοκιμάσουμε εάν λειτουργούν οι κάρτες. Τότε άρχεται μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, βλέπω κάποιους συναδέλφους ακόμα που θέλουν να ψηφίσουν. Πέρας. 34 με κάρτα και μία βουλευτής χωρίς κάρτα και θα μας λέει τι θέλει να κάνει. 35 βουλευτές και όλα καλά με τα μέλη των ομάδων. Περνάμε λοιπόν αμέσως στην έκθεση της Καρολίνε Γκρας Βαντερ Χάιντς για την διαφθορά σε τρίτες χώρες. Ε, συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. 9. Μάλιστα. Υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα από την ε, τροπολογία που είναι συμπλήρωση στην τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την 22 άρχεται η ψηφοφορία πέρας μια ψήφος παραπάνω είναι κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. ως συμπλήρωση έχουμε την 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή επίσης ως συμπλήρωση για την συμβιβαστική 8 έχουμε την 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή και στην 35 έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος καταπίπτει γιατί πέρασε η συμβιβαστική 8. Οπότε θα ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται η 35. Μετά 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική εννέα υπέρ κατά αποχές δεκτή και τελική ψηφοφορία καλό ωραία χωρί ε, ηλεκτρονικά άρχεται και πέρασε. Ε, άλλη μια ψήφος υπέρ με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια Καρολίνε. Περνάμε τώρα στο σημείο 6. Έκθεση για την συμφωνία με την Κούβα του κυρίου Μπέγκε. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Και... Πέρασε. και εσείς υπέρ. Άρα γίνεται δεκτό. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εποχές δεκτή τοπολογία 37 με διαφορετική μορφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ. Να την επαληθεύσουμε. Την 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές. Να την ξαναδούμε. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή συμβιβαστική 6 υπέρ κατά εποχές δεκτή 49 υπέρ κατά εποχές δεκτή 50 υπέρ κατά εποχές δεκτή συμβιβαστική 7 υπέρ κατά εποχές δεκτή να το ξαναδούμε. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και δικτύει, Αυτό σας είπα. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, την τελική άρχιτη ψηφοφορία. πέρας. Ευρύτατη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Μπέγκε. Και τώρα περνάμε στην ε, σύμφωνη γνώμη μία ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. τέτοιο μπέρδεμα υπάρχει εκεί σε μια μεγάλη ομάδα. Σημείο 7 ψηφίζουμε. 7. Την ε, σύμφωνη γνώμη επί της συμφωνίας. Εφτά. Σημείο 7. Για την Κούβα. απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με κτλ. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας. Και αυτό με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Σημείο 8. ψήφισμα για το σύμφωνο βιωσιμότητας υπάρχει εδώ ένα προφορικό ερώτημα. Ψηφίσμα τώρα το ψήφισμα. Στην παραγράφο 1 υπάρχει η τροπολογία 36 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές δεκτό τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές κάποιοι δεν ψήφισαν λοιπόν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και δεκτή. Ε, καλό θα ήταν να ψηφίζουν όλοι. Μετά λείπει η τροπολογία 40, καταπίπτει με συγχωρείτε η τροπολογία 40 και περνάμε συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά αποχές εδεκτή, 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά άποχες δεκτή ως πιθανή συμπλήρωση της 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 55 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58-59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 60 και 61 υπέρ κατά αποχές δεκτές 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε την υπαριθμόν 19 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή ή 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την 33 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1 και 2 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτές. 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 4 και 6 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή και ηλεκτρονικά η τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας και με μεγάλη πλειοψηφία γίνεται δεκτό συγχαρητήρια τελειώσαμε άρα με τις ψηφοφορίες και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Δεν βλέπω την εισηγήτρια όμως. so, what to do? can give me the S&D group an indication if the Μπορούν οι σοσιαλδημοκράτες να μου πούν τι γίνεται, θα ξανάρθει η συγκήτρια. So, wir fangen mal an. Wir... Ξεκινάμε. Οι φιλελεύθεροι από τη Φιλανδία ζητάνε να ξεκινήσουμε και θα του δώσουμε τον λόγο πριν από την εισηγήτρια γιατί δεν είναι εδώ. Είναι ούτως ή άλλως. Ο κύριος Τάκουλε. The floor is yours. Okay, thank you, Chair. So... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ονόματος της ΔΙΤΑ. Συμμετέχω και εγώ στην ε, Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Δεν την ακούσαμε. Βέβαια ακόμα η ΙΒΑ έχει κάνει πολλά πράγματα προκειμένου να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσιδών αξία. Η προστιθέμενη αξία τη έκθεση αυτή είναι ότι να φέρουμε μαζί τα όσα έχουν γίνει, τα όσα λειτουργούν και τα όσα μπορούν να γίνουν στο μέλλον. Υπενθυμίζοντα περισσότερο το τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο όχι τόσο με την πρόβλεψη τιμωριών και κυρώσεων, αλλά περισσότερο με μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή είναι και η προσέγγιση της εισηγήτριας. Να έχουμε δηλαδή μια καλύτερη συμμόρφωση. Ξέρετε αυτή τη στιγμή προβλέπεται δεσμευτική συμμετοχή, συμμόρφωση Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ρήτρε για την υποχρεωτική εφαρμογή τη βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλέ συναπτυσσόμενε χώρε οι οποίε δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να τηρήσουν αυτέ τι ρήτρε και αυτέ τι υποχρεώσει. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ε, πρωτοβουλίες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και στις συμφωνίες αυτές να προβλέπονται συγκεκριμένε διευκολύνσεις για τις ε, χώρες αυτές. Επίσης, στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών προβλέπονται οι δυνατότητες για ορισμένες επιχειρήσεις να αναλάβουν ε, δοντολογικές αποφάσεις, να προωθήσουν περισσότερο δηλαδή την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη και ουσιαστικά θέλουμε οι επιχειρήσεις αυτές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αν υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις να έχουν σε όλη την παγκόσμια λυσίδα αξία μια στάση ιδεοντολογική, τότε απαιτείται και απόλυτη διαφάνεια σε όλη αυτή την αλυσίδα, προκειμένου να μπορούν και οι επενδυτέ και οι να εντοπίσουν τελικά ποιες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες, οι εταιρείες εκείνες οι οποίες τηρούν τις υποχρεώσει τους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν ομοιάζουν μεταξύ τους όλες οι αλυσίδες αξίας, ούτε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ή στα πλαίσια των ίδιων δικτύων όλες οι επιχειρήσεις. Τώρα, οι επιχειρήσεις εν συνεχεία θα πρέπει να αναπτύσσουμε μία προσέγγιση η οποία να έχει να κάνει βέβαια και με τη θέση την οποία έχουν και με τη φύση της επιχείρησης, αλλά και με γενικότερες κατευθύνσεις γραμμές. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα επισήμανσης αφορά την περιβαλλοντική και κοινωνική χνηλασιμότητα, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτή τη στιγμή όμως ε, δεν καταλήγει η έκθεση σε κάποιο συμπέρασμα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε μια δεσμευτική τέτοια, υποχρεωτική τέτοια επισήμανση. Επίσης, ε, στην έκθεση αυτή γίνεται και μία αναφορά στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ως προς το ζήτημα αυτό εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς ε, οι οποίοι κατέβαλα μια κάποια προσπάθεια για να με καταλάβουν. Γιατί ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο και για μένα να διαβάζω τη σημειώσεις της συναδέλφου. Σας ευχαριστώ πάντως για την προσοχή σας. totally uh, Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι οι διερμηνείς θα μπορούσαν να μεταφράσουν και τα φιλανδοαγγλικά σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα σας ξαναδούμε σύντομα. Γεια σας. Μαρία, σειρά σου. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά οι ψηφοφορίες στις διάφορες επιτροπές ε, δυσκολεύουν τη ζωή μας. Άκουσα ένα τμήμα της παρέμβασης του συναδέλφου για το θέμα των ε, ε, αλυσίδων αξιών. Οι παγκόσμιε αλυσίδε αξία έγιναν βασικό στοιχείο τη παγκόσμια οικονομία και ακριβώ γι' αυτό ασχολούμαστε με το θέμα αυτό στην Επιτροπή ΙΝΤΑ γιατί το θέμα του εμπορίου και των επενδύσεων είναι πολύ σημαντικό στις ε, αλυσίδες ε, αξίας. Ε, η, η παραγωγή διαθώνεται γύρω από αυτές τις αλυσίδες και τις συντονίζουν ποιος οι πολυεθνικές. Ε, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για μια προσέγγιση διαφοροποιημένη ανάλογα με το είδος των επιχειρήσεων και προφανώς αυτό είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μα. Σήμερα τα τελικά προϊόντα δεν είναι παρά το 25% του παγκόσμιου εμπορίου. Ε, αυτό δείχνει σε ποιο βαθμό το να ασχοληθούμε με τις αλυσίδε αξία είναι σημαντικό. Ως πρώτος ε, εισαγωγέας και εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμπορική τη πολιτική για να την καταστήσει μοχλό, ούτω ώστε αυτέ οι αλυσίδε να εξυπηρετήσουν την βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλου και να συνεισφέρει σε μια πιο δίκαιη παγκοσμιοποίηση. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένω με την Επίτροπο Μάλστρομ. Δηλαδή ότι το εμπόριο θα πρέπει να είναι δίκαιο εμπόριο και να μην αποκλεί κανένα και η παγκοσμιοποίηση να μην αφήνει κάποιου στο περιθώριο. Ε, ε, μιλάμε για, για την χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης και η Κομισιόν θέλει ε, μια προοδευτική στάση ε, που να βασίζεται σε κανόνες, διαφάνεια, υπευθυνότητα, εταιρική ευθύνη, σεβασμό των εταιρικών κανόνων και κοινωνικών κανόνων. Αυτός ο προβληματισμός έγινε μέσα στα πλαίσια όπου η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική έγινε βασικό διακύβευμα και έχει τεράστιο Δηλαδή, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον οι πολίτε για αυτό το θέμα. Μας ε, μιλάνε για τις ανησυχίες του. Θέλουν μια πιο δίκαιη και πιο διαφανή εμπορική πολιτική. Προηγουμένω μίλησαμε για το θέμα της εκμελασιμότητας, αλλά πιο δημοκρατική, πιο δίκαιη και ε, σε φάση με τις προκλήσεις τη εποχής μας, δηλαδή πολέμηση των ανισοτήτων, ε, την κλιματική αλλαγή, τη φοροδιαφυγή. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό σε αυτή την ευθύνη να μιλήσουμε για την ε, εταιρική ευθύνη, για τη διαφάνεια και την ε, κοινωνική ευθύνη, την ε, φορολογική ευθύνη και την παραγωγική ευθύνη. γιατί η Ευρώπη των αξιών που υπερασπιζόμαστε θα πρέπει να υπάρχει και στο διεθνές εμπόριο και το θέμα εδώ δεν είναι μόνο θέμα αρχών, είναι αυτό το εμπόριο μια πραγματική προστιθέμενη αξία. Αυτή η έκθεση φυσικά έχει όλες αυτές τις προτεραιότητες, δεν πρόκειται σήμερα τώρα να κλείσω αυτή τη συζήτηση. Αντίθετα, μόλις ξεκινάει η συζήτηση και φυσικά θα είμαι προσεκτική. Άκουσα τις ανησυχίες του Άλντε για μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Ε, υπάρχει επίσης και το θέμα των εντάσεων ανάμεσα στην, στο τι είναι υποχρεωτικό και την εθελοντικό. Αυτά τα συζητήσαμε όταν συζητήσαμε τα μεταλλεύματα από εμπόλεμες περιοχές. Ε, κάποια στιγμή πιστήκαμε ότι χρειάζεται μια ευελιξία στις προτεραιότητες. Ελπίζω να έχουμε και, την, εδώ την ίδια προσέγγιση, να βρούμε δηλαδή μία λύση που θα επιτρέπει να απαντρέψουμε και τις αξίες που τις θέλουμε, τις επασπιζόμαστε και από την άλλη μία σημαντική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ε, στις παγκόσμιες αυτές αλυσίδες ε, αξιών. Ευχαριστώ. Και τώρα σκιώδεις εισηγητές. Αυτό το πρώτα. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης της, για το, τις αλυσίδες αυτές. Ε, θα μας απασχολήσει και μας απασχόλησε και στις 20 Μαρτίου. Θα θυμάστε τις παρατηρήσεις που είχε κάνει ο κύριος Βαλέζα εν ονόματί μου τότε. η συμπερίληψη των δικαιωμάτων των παιδιών που δεν, υπάρχουν, δεν υπήρχαν πριν και η συμπερίληψη των μικροεπιχειρήσεων και η αναφορά στις ειδικές, στα ειδικά χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία πριν, τώρα υπάρχουν. Μια άλλη πρόταση κάναμε επίση αλλά δεν ε, ληφθεί υπόψη. Και ακριβώ γι' αυτό θα καταθέσουμε τροπολογίε. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω όμω για αυτά. Θέλω να μιλήσω για το περιεχόμενο της ε, έκθεση και να σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχά. την ε, υποχρεωτική πρώτερη άδεια. Σε προηγούμενες εκθέσεις του Κοινοβουλίου υπήρχε μία συνενετική θέση. Παραδείγματος χάρη όσα ε, ο, το, ο ILO είχαν μια κοινή θέση. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να βρούμε μια συνένεση για αυτό το πολύ σημαντικό σημείο. Νομίζω ότι σε η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ είναι πάρα πολύ σημαντική, ε, σημαντικός είναι όλος και του ΟΣΑ, καθώς και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στα διεθνή φόρουμ, ούτως ώστε να υπάρξει μια πολυμερής πρόοδο και να υπάρχει και ένα δίκαιο και υπεύθυνο εμπόριο για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και των καταναλωτών. Δέκα από τις 12 χώρες που υιοθέτησαν τα εθνικά σχέδια δράσης για τις αρχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, από αυτές τις 10 χώρες, τα, οι 8 είναι μέλος, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Κομισιόν πρέπει να μας ετοιμάσει μια ανακοίνωση για αυτά τα θέματα. Ε, πολύ λεπτομέρη. Και εμείς πρέπει να κάνουμε μια δική μας, ένα δικό μας προβληματισμό. Και επιπλέον θέλω να σταθώ πριν κλείσω στο σημείο των μικροεπιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων πώς θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά του, γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, ούτε τους ανθρώπινους πόρους που έχουν οι, πολλοί εθνικές. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό το σημείο, γιατί και αυτές οι επιχειρήσεις ε, συμμετέχουν στις ε, αλυσίδες αξιών. Επίσης, υπάρχουν τα θέματα των ένδικων μέσων για πολίτες τρίτων χωρών εναντίον επιχειρήσεων ε, που προέρχονται από ένα κράτος μέλος. Ε, μιλάμε για μία πρόταση που θα πρέπει να γίνει για το σημείο 13, ούτως ώστε να ξεκινήσει μία, ένας προβληματισμός για τους κανόνες ανταγωνισμού. Το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και νομικά και οικονομικά και θα πρέπει να το συζητήσουμε και σε επίπεδο ΩΣΑ ή επίπεδο ΙΕ, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως πρέπει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο σε όλα αυτά τα θέματα, ειδικά για τα ένδικα μέσα. και το Συμβούλιο το είπε στις 12 Μαΐου στα συμπεράσματά του και το Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε αυτή την ιδέα, την ιδέα της εταιρική ευθύνη σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε τρίτες χώρες. Εκεί είχαμε ζητήσει να γίνει πλέον προβληματισμός για αυτό το θέμα. Όταν ε, χτίζουμε ένα σπίτι δεν το χτίζουμε από την ε, στέγη, αλλά από τα θεμέλια. Για να έχουμε αποτελεσματικούς νόμους θα πρέπει να ξεκινήσουμε από, τα, από τη βάση, να ξεκινήσει μια διαδικασία προβληματισμού, ενδελεχής, ε, με διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων μερών, με όλες τις αρχές και τους φορείς και να λάβουμε υπόψη μας το ύψιστο συμφέρον των πολιτών. Αυτή την προσπάθεια ε, θα πρέπει να την ξεκινήσουμε στο Κοινοβούλιο με μελέτες, με σεμινάρια, με ακροάσεις, ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι stakeholders. Είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να καταλήξει σε έναν οδικό χάρτη. Γιατί μιλάμε για ένα ε, περίπλοκο νομικό πλαίσιο. Κλείνω συγχαίροντα την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. Θέλω να τη πω ότι είμαστε στη διάθεσή τη. Ε, έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κανείς άλλος από τους πιο δυσηγητές δεν είναι παρόν. Δύο ακόμα συνάδελφοι όμως θέλουν να πάρουν το λόγο. Α, συγγνώμη. Αν Μαριμινέρη είστε εδώ πέρα. Αλλά έβλεπα το όνομα του κυρίου Ζαντό, γι' αυτό δεν σας είδα. Απόλυτη σύγχυση κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρένα για την δουλειά της την έκθεση την κυρία Αρένα Έχουμε δύο κατευθύνσεις τώρα, η μία πηγαίνει προς περισσότερο κέρδος ε, λιγότερους κανόνες, ενώ οι άλλοι θέλουν να κερδίσουν όλοι από το εμπόριο. Η έκθεση αυτή επιλέγει λοιπόν την δεύτερη κατεύθυνση και δεν ε, ξεχνάει τη σημασία της υγιούς οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν τη μεγάλη της σημασία ε, και έχει μεγάλη σημασία να φροντίσουμε να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Λέει βεβαίως πως η κυρία Ρένα πως ε, θα πρέπει να περάσουμε από το εθελοντικό στο υποχρεωτικό επίπεδο του ΟΗΕ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα μέτρα που προτείνονται ε, για υποχρεωτικές ρήτρες ε, στις ε, εμπορικές συμφωνίες, ρήτρες standstill με κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενημερωθούν και οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος που αδιαφορεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι πολύ ικανοποιημένη λοιπόν με αυτή την έκθεση και ε, θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, Χάιντι Χάουταλα. Um, uh, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω το σχέδιο έκθεσης αποτελεί πολύ σημαντική συμβολή στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Εμπόριο για όλους», «Trade for All» που όπως μας λέει και η Μαρία Ρένα βασίζεται στις αξίες, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που η συγγήτρια τονίζει στην έκθεση αυτή ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού προκειμένου να αποφύγουμε οι πιο υπεύθυνε επιχειρήσεις να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, μόνο και μόνο επειδή ακολουθούν επιστά τους κανόνες. Επειδή δεν παραβιάζουν τους κανόνες, δεν καταπατούν δικαιώματα και δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Αυτή τη λογική λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα πρέπει να προωθούμε περισσότερο τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτές να επιβραβεύουμε και όχι τις άλλες. Θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση που να βασίζεται στη δέουσα επιμέλεια, όπου να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία να είναι εκτελεστά και δεσμευτικά, και όχι μόνο η Γαλλία αλλά και άλλα κράτη-μέλη. Μην το ξεχνάμε, έχουν εθνικέ νομοθεσίες οι οποίες είναι πολύ θετικές και νομίζω ότι οφείλουμε και οι υπόλοιποι να συμβάλλουμε για να δημιουργήσουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι ανάλογο. Θα ήθελα τώρα να επιστήσω την προσοχή σας στην παράγραφο 12 της έκθεσης που καλεί τα κράτη-μέλη να γνωστοποιήσουν στο κοινό κατόπιν αιτήματο τα τελωνιακά στοιχεία που συλλέγονται από μέρη τα οποία εμπορεύονται προϊόντα αγαθά που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι είναι ένας συνεχής αγώνας που δίδεται για πάρα πολύ καιρό τώρα προκειμένου να μπορούν οι ε, τελωνιακές αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τα δεδομένα τα οποία συσσωρεύονται σε εθνικό επίπεδο μόνο αυτή τη στιγμή. Αυτό θα αποτελούσε μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να γνωρίζουμε καλύτερα την πραγματική προέλευση των προϊόντων. Νομίζω λοιπόν στο κεφάλαιο αυτό θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πρόοδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάταξη αυτή να παραμείνει στο σχέδιο έκθεση. Τώρα η πολιτική μου ομάδα θα ήθελε να προσθέσει στην έκθεση αυτή κάποια στοιχεία να επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο καταρχάς το πεδίο εφαρμογής των συστάσεων αυτών που να καλύπτουν πλέον όχι μόνο το εμπόριο αλλά και τις επενδύσεις. Επίσης, θα θέλαμε το σύστημα GSP Plus για το, τις γενικευμένες προτιμήσεις, καθώς επίσης και για τα εμπορικά ωφέλη να αναπτυχθεί λίγο περισσότερο στην έκθεση και ως προς αυτός νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε λίγο περισσότερο τις ζώνες επεξεργασίας των εξαγωγών. Μήπως θα έπρεπε οι ζώνες αυτές να αποκλειστούν από την επιβολή δασμών στα πλαίσια του GSP+. Αυτό θα ήταν μια πρόταση της δικής μου πολιτικής ομάδας. Πάντως προσβλέπω και στη μελλοντική συζήτηση που θα έχουμε για την επεξεργασία της έκθεσης αυτής. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο έκθεσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Κοιτώντας την ιδεολογική έκθεση, βλέπω ότι η εισηγήτρια λέει ότι πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνεται για την εμπορική της πολιτική. Άρα πρέπει να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όντως η εμπορική μας πολιτική μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το εξηγεί πολύ καλά η εισηγήτρια, η οποία αναφέρεται επίσης και στην ανακοίνωση Trade for All, εμπόριο για όλους. Στα πλαίσια τη πρωτοβουλίας αυτής λέγεται ότι χρειαζόμαστε υπεύθυνε αλυσίδες αξία. Πώς μπορεί όμω να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να θίξουμε τρία βασικά σημεία, θεωρώ, για να οριοθετήσουμε, να πλαισιώσουμε και λίγο τη συζήτηση με τις παγκόσμιες αλυσίδε αξίες να φερόμαστε βασικά σε εμπορικές δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αναγκαστικά στο στερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, οι αλυσίδες αυτές αξίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες, καλύπτουν ε, απλά μέχρι πολύ πολύπλοκα προϊόντα και τρίτον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αποφύγουμε ανεπιθύμητες επιπτώσεις από την πρωτοβουλία μας αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να καταστρέψουμε θέσεις απασχόλησης, θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Έχοντας λοιπόν αυτά κατά νου, βλέπουμε ότι η έκθεση καλύπτει πάρα πολλά ζητήματα, καλύπτει από διάφορες σκοπιές και οπτικές γωνίες της παγκόσμιας αλυσίδας αξίες, αναφέρεται στην επισήμανση των προϊόντων, αναφέρεται στην ευθύνη των κυβερνήσεων όσον αφορά τι συμφωνίε δεύτερων συναλλαγών, όσον αφορά το σύστημα GSP+, αναφέρεται στη δέουσα επιμέλεια, αναφέρεται επίσης και στη διεθνή διάσταση όταν μιλάει για την πολυμέρεια, την πολυμερή προσέγγιση απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα αυτό και ότι καλούμεθα να αναλάβουμε δράση σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Εγώ εκπροσωπώντας τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου μιλάω για τα εμπορικά ζητήματα, αλλά εμπλέκονται και πολλές άλλες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζετε. Η εμπορική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προς αυτό το σχέδιο έκθεσης προσπαθεί να πλαισιώσει την εμπορική πολιτική στα πλαίσια της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ θα πρόσθετα και άλλες πολιτικές όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει να είμαστε πιο συνεκτικοί με την περιβαλλοντική πολιτική, με την εξωτερική πολιτική και με πολλές άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια λοιπόν των περιορισμών και των αρμοδιοτήτων της εμπορικής πολιτικής τώρα, πολλά σχόλια θα μπορούσε να κάνει κανείς. Δεν θα ήθελα να επισέλθω αυτή τη στιγμή σε κάθε σημείο ξεχωριστά. Ορισμένες παρατηρήσεις γίνανε ήδη από κάποιους ευρωβουλευτές. Ενδεχομένως λοιπόν να αφαιρθώ στι παρατηρήσεις αυτές στην παρέμβασή μου. ένα ευρωβουλευτή αναφέρθηκε στο DSD, στο κεφάλαιο αυτό που έχει να κάνει με τη δέουσα επιμέλεια, καθώς επίσης και με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και στις ρήτρες standstill, στο ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να πετύχουμε. Ακρογωνιαίος λήθος της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαπραγματεύση διμερών συμφωνιών είναι να καταφέρουμε να προωθούμε τα διεθνή πρότυπα, τα διεθνή αυτά πρότυπα, όπως για παράδειγμα η Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θέτουν τελικά τη βάση το κριτήριο εκείνο το οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα πρέπει να συμμορφωθούν και οι υπόλοιπε χώρες. Σε ζητήματα όπως το CSR, αν θα πρέπει η κοινωνική εταιρική ευθύνη να είναι υποχρεωτική ή εθελοντική. Πολλά και στο παρελθόν συζητήσαμε το ζήτημα αυτό. Η προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα εργαλεία για την αξιολόγηση τη κοινωνική εταιρική ευθύνη, που πιστεύουμε εμεί ότι θα πρέπει όμω να μείνει εθελοντική. Συνεχίζεται όμω η συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Ξέρετε ότι έχουμε και το έγγραφο προβληματισμού για τη χαλινακόγηση τη παγκοσμιοποίηση και εκεί θίγουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και περιμένουμε και τι δικέ σα τι παρατηρήσει. Κάποια άλλα ζητήματα τώρα. Κανονισμό Βρυξέλλε 1. Καταγράφω τι παρατηρήσει που έγιναν προ αυτό. Δεν είμαι ειδήμων για το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Καταγράφω πάντω τι παρατηρήσει και τι ιδέε σα και το ότι θέλετε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα τελωνιακά δεδομένα. Αυτό είναι έκκληση περισσότερο προ τα κράτη-μέλη, βέβαια, έτσι δεν είναι. Ε, προκύπτουν κάποια ζητήματα όσον αφορά το εμπορικό απόρριτο, στι δραστηριότητε κάποιων επιχειρήσεων και αυτό όμω θα το εξετάσουμε περαιτέρω. Μια σημαντική πτυχή τώρα της, του ζητήματος που εξετάζουμε το έθεσε και η εισηγήτρια ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του κεφαλαίου DSD. Είναι δεσμευτικός ο χαρακτήρας των ρητρών αυτών για τους εταίρους μας, ότι δεν προβλέπονται κυρώσεις. Εμείς προσπαθούμε πάντως να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις αυτές για να προωθήσουμε τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και μια πρόσφατη εξέλιξη που είχαμε στην Κεντρική Αμερική. Είχαμε την πρώτη διάσκεψη στην περιοχή αυτή για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στις αρχές Μαΐου. Η διάσκεψη αυτή ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, συμμετείχε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και ο ΩΣΑ, καθώς επίσης και ο ιδιωτικός τομέας. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι πολλές συζητήσει δεν είχαν να κάνουν μόνο με κάποια βασικά προϊόντα, γιατί ξέρετε πολύ συχνά όταν μιλάμε για παγκόσμιες αλυσίδες αξία, οι περισσότεροι νομίζουν ότι μιλάμε για είδη ένδυσης ε, ή για τα γεωργικά προϊόντα. Θίξαμε όμως και πολλούς άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα το τομέα των φαρμάκων ή τον τομέα της πληροφορικής και τα σχετικά ψηφιακά προϊόντα και οι παρατηρήσει που είχαμε ήταν ιδιαίτερα θετικέ όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Η βασική μα ανησυχία δεν είχε να κάνει τόσο πολύ με τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα τη εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά περισσότερο το ζήτημα τη χρηματοδότηση. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να θίξουμε, διότι επηρεάζει πολλέ από τι προτάσει τη έκθεση, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την προώθηση, την επιβολή υποχρεώσεων έξωθεν προς επιχειρήσεις οι οποίες δεν υφίστανται, δεν έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική μας πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να νομοθετήσουμε μέσω αυτής στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιβάλλουμε εμείς κανόνες σε εξωτερικέ επιχειρήσει με τον ίδιο τρόπο που επιβάλλουμε σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσουμε να θίξουμε τα, όλα αυτά τα ζητήματα στους συναδέλφους εκείνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται και αυτοί στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Ένα ακόμα στοιχείο που πιστεύω ότι θα μπορούσε να τονιστεί περισσότερο στην έκθεση είναι ο ρόλος των καταναλωτών. Οι καταναλωτέ μπορούν και αυτοί να επηρεάσουν τα πράγματα με τι επιλογέ που κάνουν, μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια των παγκόσμιων αλυσιδών αξία. Και ολοκληρώνοντα να πω ότι συμμεριζόμαστε κοινού στόχου. Βλέπουμε ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει εδώ πέρα η συγγήτρια, να γίνουν οι αλυσίδες αυτές αξίας πιο διαφανείς και να εξυπηρετούν τελικά την αηφόρο ανάπτυξη. Η δική μας η προσέγγιση μπορεί μερικές φορές να διαφοροποιείται σε κάποια σημεία, μπορεί να, να μην συμφωνούμε στα πάντα, για συγκεκριμένα ζητήματα μπορεί να διείστανται οι απόψεις μας, αλλά εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο αυτό που έχουμε μαζί σας και εν τέλει να πω ότι η εισηγήτρια είπε πολύ σωστά ότι βρισκόμαστε απλώ στην αρχή τη συζήτηση. Δεν ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση. Πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε μακροπρόθεσμα. Τα ζητήματα αυτά είναι μία νυχτή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διευθετηθούν. Θα πετυχθεί χρόνο. Αυτό που ελπίζουμε να δούμε είναι την πιο έντονη εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων στον τομέα αυτό. Προσθέτουμε λοιπόν στη συνέχιση του, του διαλόγου. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες και παρεμβάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Για την αναφορά στον ΟΗΕ, στον ΩΣΑ και στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, δουλέψαμε από αυτού. Αντί να, δουλέψουμε, ε, να φτιάξουμε νέες αναφορές ε, που θα βρίσκει, δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους, το να δουλεύουμε τους κλασικούς φορείς όπως τον ΟΗΕ και τον ΩΣΑ και τον ILO ε, είναι η κλασική φορής αναφοράς ε, και δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε έτσι νέα πρότυπα. Οι επιχειρήσεις δουλεύουν ήδη με αυτά. Είναι σημαντικό να το πούμε. Και στο ΝΟΣΑ, όταν μιλάμε για τη δέουσα επιμέλεια, μην ξεχνάτε ότι εκεί λαμβάνουμε υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές επιχειρήσεις. Άλλο μία μικρομεσαία επιχείρηση, άλλο μία πολυεθνική. Η προσέγγιση διαφοροποιείται ανάλογα με το είδο επιχείρηση. Σημαντικό αυτό. Όταν μιλάμε για την δεύτερη επιμέλεια στα πλαίσια των λυσίδων αξιών, ε, στην πραγματικότητα μιλάμε για διαφάνεια τελικά. Έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να είχαμε κάνει πριν από λίγα χρόνια. Δεν με είχαν εκλέξει ακόμα σε ό,τι αφορά την εναρμονισμένη, ε, τα εναρμονισμένα λογιστικά των επιχειρήσεων. Σήμερα δεν υπάρχει επιχείρηση, επιχείρηση χωρίς τέτοια ε, λογιστικά. Ε, Κανένα δεν θα επένδυσε σε μια επιχείρηση που δεν είχε αυτή την αρμονισμένη ε, λογιστική, γιατί δεν θα είχε την ασφάλεια. Εδώ μιλάμε επίση για το ρόλο των καταναλωτών. Συμφωνώ ότι ο καταναλωτή ε, σίγουρα έχει ένα ρόλο και μια ευθύνη στο τέλο όμω, στην άκρη τη αλυσίδα. Αν δεν του εγγυηθούμε όμω μια τυποποιημένη προσέγγιση, διαφανή προσέγγιση, σε σχέση με το τι περιέχει αυτή η αλυσίδα, πώ θα παίξει το ρόλο του υπεύθυνου καταναλωτή. Η δέουσα επιμέλεια αυτό εξασφαλίζει. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή σε έναν υπεύθυνο καταναλωτή να κάνει μια υπεύθυνη κατανάλωση με τις απαραίτητες ε, τυποποιημένες πληροφορίες, όσο περισσότερο τυποποιημένες γίνεται σε αλυσίδες αξιών που είναι παγκόσμιες. Τώρα αυτό αφορά τις, ε, επιχει... τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή τις ξένες. Φυσικά δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε για τις ξένες επιχειρήσεις, αλλά πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι τμήμα αυτών των αλυσίδων αξιών και μπορούμε λοιπόν να τους επιβάλλουμε κάποια πράγματα ακόμη και όταν αρσιοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ναι, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος, να προάγει τις αξίες. Ε, και εδώ δεν μιλάω μόνο για την οικονομική αξία που παράγουν οι λυσίδες αξιών, αλλά και για την ανθρώπινη αξία Είπατε προηγουμένω ότι δεν μπορούμε να καταστρέφουμε θέσει απασχόληση. Σωστό. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να καταστρέφουμε θέσει απασχόληση. Αλλά ούτε είμαστε εδώ για να καταστρέφουμε ζωέ. Εάν πρέπει να δημιουργηθεί μία ε, θέση απασχόληση, και αν το δεχόμαστε αυτό, πολλό δε μάλλον η ανθρώπινη ζωή. Αυτό το νόημα έχει και η αλυσίδα αξία και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, Κάνοντα βεβαίω του απαραίτητου συμβιβασμού. Σα ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Να σας πω ότι δεδομένου του περιορισμού στις σελίδες που έχουν αυτές οι εκθέσεις και εγώ ακόμα η ίδια θα υποβάλω τροπολογίες. Άρα οι δικές σας τροπολογίες εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτες. Προφανώς το περίμενα. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε το σημείο 9. 6 Ιουνίου για τις τροπολογίες. Στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. 10 και 11 Ιουλίου. Επόμενο σημείο. Το αγαπημένο μου. Τα διάφορα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε στο 11. Η επόμενης επόμενη 19 και 20 Ιουνίου είναι αυτές οι ημερομηνίες. Αυτά. Γεια σας.